Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie Platz. Καθίστε παρακαλώ συνάδελφοι. Και ξεκινάμε. Έχετε λάβει την ημερήσια διάταξη. Την έχετε μπροστά σα. Το πρώτο. Λοιπόν, ζήτημα είναι κατά πόσο εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αντιρρήσεις κατά του σχεδίου ημερήσιας διάταξης. Όχι. Ως εκ τούτου εγκρίνεται η μυρική διάταξη, όσο έχει. Και περνάμε στο 2. Ανακοινώσει του Πρόεδρου. Μία συνηθισμένη ανακοίνωση. Στο διαδίκτυο ζωντανά αναμεταδίδεται η συνεδρίασή μας. Να το έχετε υπόψη σας και άρα να μιλάτε και με σωστό ρυθμό για να σας παρακολουθούν και διερμηνήσει. Κατά δεύτερον, μία, ένα κατάλογο επιστολών έχετε μπροστά σας που σας έχει αποστείλει η γραμματεία. Αν θέλετε να δείτε τι επιστολές αυτέ, είναι στη διάθεσή σας η γραμματεία για να σας βοηθήσει. Για τις διαπραγματευσεις ενα έναμπτος ε, γύρος 16-22 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται και, και δέκατος γύρω πριν από τη διάσκεψη του Ναϊρόμπι, το Δεκέμβριο. Ίσως ε, λοιπόν μπορούμε να αναμένουμε κάποιες ε, πρόοδους σε αυτό το πλαίσιο. Πριν ε, επίσημα ξεκινήσουμε και τις συνεδρίες τα θέματα, να σας υπενθυμίσω, το έκανα και ηλεκτρονικά άλλωστε, ότι μια καλή φίλη της Επιτροπής μας, η Λένα Ικ, πριν από 10 ημέρες απεβίωσε πριν από 10 μέρες, στις 10 Σεπτεμβρίου. Πολλοί τη γνώριζαν καλά, τη Λένα X, και ήταν εντυπωσιασμένοι από από την εργασία της, από τη δουλειά της και είμαι ιδιαίτερα λυπημένος για την ε, είδηση αυτή που λάβαμε ιδιαίτερως επειδή ήταν μόνο 28 χρονών. Και η κηδεία έγινε στις Βερσαλίες. Σίγουρα θα τη θυμόμαστε και θα θυμόμαστε πάντα και την δημιουργική της δουλειά και το δημιουργικό της έργο. Σας ευχαριστώ. Να περάσουμε στο 3 έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης, των τελευταίων συνεδριάσεων. Ούτε εδώ έχω λάβει παρατηρήσεις. Αν μέχρι τα τέλη της συνεδρίασης δεν εκφραστούν ενστάσεις, θα θεωρήσουμε ως συνήθως ότι τα πρακτικά εγκρίνονται. Και τώρα περνάμε στο 4 της σημερινή διάταξης και χαίρομαι ιδιαίτερος που έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Γενικής ε, Διεύθυνσης Εμπορίου, το Μάουρο Πετριτσιόνε, προκειμένου να συζητήσουμε και μαζί του τη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα νέο σύστημα προστασίας ε, επενδύσεων σε εμπορικές ε, συμφωνίες και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη συμφωνία TTIP. Θα ήθελα παρά αυτό να του δώσω το λόγο προκειμένου να ξέρουμε ε, πιο επακριβώς το τι προτείνεται. Σας παρακαλώ λοιπόν, να πάρετε λόγο. Thank you very much, Mr. Chairman. Ε, very happy. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που επανήλθα στην Επιτροπή σας για να σας δώσω κάποιες πρώτες ε, σκέψεις για τις προθέσεις της Κομισιόν για την πρόταση προς τη ΣΥΠΑ για την προστασία των επενδυτών και την επίλυση διαφορών επενδυτών. Η Επίτροπος ομάδα των θα ήθελε να είναι παρούσα σήμερα, αλλά βρίσκεται στις Ηνωμένε Πολιτείε για συζητήσεις. Θα σας εξηγήσει η ίδια γιατί κάναμε την επιλογή αυτή ωστόσο. Ξεκινώ, Πρόεδρε, με δύο λόγια για τη διαδικασία. Πρόκειται για μια κατά κάποιο τρόπο άνευ προηγουμένου διαδικασία. Δεν είναι επίσημο το κείμενο, είναι σχέδιο της Επιτροπής. Το στείλαμε, το μεταβιβάσαμε στο Συμβούλιο ταυτόχρονα με το Κοινοβούλιο και θα ξεκινήσουμε τη συζητήση μας στο Συμβούλιο όπως ήθιστε πριν η πρόταση μετατροπή σε επίσημη πρόταση που θα υποβάλει η Ένωση στη ΣΥΠΑ στις διαπραγματεύσεις. Μερικές φορές η Επιτροπή έχει εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις για την πρόταση αυτή, αλλά όχι συχνά. Προφανώς αυτό είναι μια πολύ ειδική περίπτωση. Είναι θέμα εξαιρετικής σημασίας ε, που δημιούργησε εξαιρετικές συζητήσεις. Στόχος μου σήμερα πάντως είναι να σας ε, παρουσιάσω την πρόταση, να απαντήσω σε ερωτήσεις που έχετε στο μέτρο του δυνατού, να φροντίσω να απαντηθούν όσες δεν μπορώ να απαντήσω σήμερα, το σύντομο του δυνατό δηλαδή, και να δούμε πώς εξελιχθεί η συζήτηση. Επίσης η Επιτροπή δημοσιοποίησε το σχέδιο αυτό και αυτό είναι μια πρωτοφανής περίπτωση. Συνήθως δεν δημοσιοποιούμε σχέδια κειμένου. Όπως ξέρετε δημοσιοποίησαμε τις προτάσεις που κάνουμε στις διαπραγματεύσεις Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για τους λόγους που προανέφερα και πάλι, αποφασίσαμε ότι δεν ήταν σκόπιμο να περιμένουμε και αποφασίσαμε να κοινοποιήσουμε το σχέδιο. Πρόεδρε, το θέμα το συζητούμε 1,5 χρόνο και. Η προσπάθεια να υλοποιήσουμε την δέσμευση της Θείας Μάλστρομ στο ξεκίνημα της θητείας ότι θα χρησιμοποιήσουμε το TTIP ως ευκαιρία για μια σε βάθος μεταρρύθμιση του συστήματος προστασίας των επενδυτών και επίλυσης διαφορών με επενδυτές. Ξέρουμε πόσο ένταση έχει η σχετική συζήτηση. Αυτό που κατέστη ωστόσο σαφές, ανεξάρτητα από την πλευρά με την οποία είναι κάποιος, είναι ότι υπήρχε γενικευμένη έλλειψη εμπιστοσύνη των πολιτών στο σύστημα διατησίας που προκύπτει από την εμπορική, τη διαδικασία εμπορικής διατησίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ένα σαφές μήνυμα που βγήκε και το Κοινοβούλιο σαφώς το ερμήνευσε ε, αυτό ως πραγματική επιθυμία ήταν ότι έπρεπε να προχωρήσουμε προς ένα περισσότερο δικαστικού χαρακτήρα σύστημα για την επίλυση διαφόρων με επενδυτές. Το Μάιο ετοιμάσαμε ένα concept paper που συζητήθηκε και εδώ. Το κείμενο παρακολουθεί πιστά τη δομή και τους στόχους του κειμένου εκείνου. Δύο βασικά στοιχεία περιέχονται εδώ. Πρώτον, προστασία των επενδύσεων. Η ολοκλήρωση δηλαδή του έργου που έγινε με την υφιστάμενη προσέγγιση της επιτροπή μετά την συνθήκη τη Λισαβόνα, εξασφαλίζοντα ότι τα πρότυπα προστασία των επενδύσεων ε, είναι σαφή, καλά καθορισμένα, λειτουργικά, μπορούν να αποφασιστούν σε δικαστήριο και, πιο σημαντικό, δεν επηρεάζουν το δικαίωμα των κυβερνήσεων να ρυθμίζουν νομοθετικά προς όφελος του, ε, της κοινή ωφέλεια, του δημόσιου ωφέλους. Το δεύτερο δεδομένο ήταν να προχωρήσουμε από ένα σύστημα ιδιωτικής δικαιοσύνης που είχε κρυθεί απαράδεκτο ένα σύστημα δημόσιας δικαιοσύνης όπου το ζήτημα λύνεται από ένα σώμα επαγγελματιών δικαστών που έχουν τα στοιχεία για να παράσχουν στον πολίτη εμπιστοσύνη, βεβαιότητα στην αμεροληψία, ικανότητα και σωστή δουλειά. Not surprisingly, these are exactly the requirements that uh, the Φαντάζομαι ότι δεν σα εκπλήσει πω αυτά ακριβώς ήταν τα αιτήματα του Κοινοβουλίου στο ψήφισμά σα για το TIP. Βελτίωση του επίπεδου προστασία σε ασφαλέ ε, νομικό επίπεδο, ε, δικαίωμα, τι αναφορά στο δικαίωμα ρύθμιση των κρατών και νέο σύστημα για ένα σύστημα επίλυσης επενδυτικών διαφορών με διαφάνεια, ανεξαρτησία, επαγγελματισμό από δημόσια τοποθετημένου δικαστέ με μια διαδικασία προσβάσιμη στο κοινό και ακόμα πιο σημαντικό με τη δυνατότητα ένδικου μέσου για την διόρθωση οποιοδήποτε σφάλματος στην απονομή δικαιοσύνη σε πρώτο βαθμό. Τώρα να σας πω πως το κάναμε εντάχει. Το κύριο νέο στοιχείο στην πρόταση αυτή είναι ένα νέο άρθρο για το δικαίωμα νομοθετικής ρύθμισης με τίτλο επενδύσεις και κανονιστικά μέτρα. Ξεκινά αναφέροντας ρητά το δικαίωμα, ότι το δικαίωμα νομοθετικής ρύθμισης για δημόσιες πολιτικές διαφυλάσσεται απολύτως. Επίσης, στη διάταξη γίνεται σαφές ότι οι, επενδυ... οι διατάξεις για την προστασία των επενδύσεων δεν εμποδίζουν τις κυβερνήσεις ε, να αλλάξουν το νομικό πλαίσιο ακόμα και αν τέτοιες αλλαγές μπορεί να επηρεάσουν αντικά της επενδύσεις. Αυτό που οι εμπειρογνώμες αποκαλούν ως ρήτρα μη σταθεροποίησης. Αυτό χρειά, προέκυψε στις δημόσιες συζητήσεις όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα πρότυπα προστασίας για, για την ισότιμη προστασία αλλά και για την έμεση προστασία. Πήγαμε και ένα βήμα παραπέρα. Αντί να πειράξουμε περισσότερο το ίδιο το πρότυπο, το επίπεδο, θέσαμε στο άρθρο το ίδιο το άρθρο μια τέτοια διάταξη που εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα προστασίας. Το δεύτερο στοιχείο αφορά τον τρόπο επίλυσης ε, διαφορών για τις επενδύσεις. Θα υπάρχει ένα σύστημα δικαστήριων επενδύσεων με πρώτο βαθμό, με πρωτοβάθμιο δικαστήριο με 15 δικαστές και ένα κατέφεση δικαστήριο με 6 μόνιμους δικαστές που ορίζονται δημοσία. Στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο οι 15 δικαστές θα ορίζονται από κοινού για 6 χρόνια από την Ένωση και τη ΣΥΠΑ και θα είναι οι μόνοι που θα δικαιούνται να κρίνουν διαφορές για επενδύσεις βάσει του TTIP. Με την θέση ισχύ θα, τεθεί, θα ξεκινήσει η τοποθέτηση. Πέντε θα είναι πολίτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέντε πολίτες των ΗΠΑ και πέντε από τρίτες χώρες. Κάθε πλευρά θα επιλέξει τους δικαστές της δικής του ηθαγένειας. Εμείς αποφασίσουμε ποια διαδικασία θα ακολουθήσουμε. Για τους εκπροσώπους τρίτων χωρών θα το συζητήσουμε με τη ΣΥΠΑ για να συμφωνήσουμε επί μιας διαδικασίας επιλογής. Αυτό δεν είναι τόσο σύνθετο όσο νομίζετε, γιατί υπάρχουν αντίστοιχες ρυθμίσει στα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα και για το είναι όργανο για το εφετείο. Εμείς είμαστε ενεργοί, ενεργά μέλη στις, και οι Ηνωμένε Πολιτείε σε αντίστοιχα τέτοια όργανα, οπότε μπορούμε να βρούμε τρόπους επιλογής των ατόμων με τα αναγκαία χαρακτηριστικά. Οι δικαστές θα πρέπει να έχουν πολύ ψηλά, επίπεδο, πολύ ψηλά προσόντα, αντίστοιχα με αυτά που απαιτούνται για μέλη διεθνών, μόνιμων διεθνών δικαστηρίων οι διαφορές βάσει του TTIP θα ανατίθενται τυχαία με ένα μηχανισμό επιλογής ε, τριών δικαστών που θα δικάζουν μια συγκεκριμένη διαφορά. Ένας Ευρωπαίος, ένας Αμερικανός και ένας τρίτος από τρίτη χώρα. Η επιλογή θα γίνεται απόλυτα τυχαία. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου που θα ανήκει σε τρίτη χώρα θα έχει ρόλο διαχείριση του συστήματος, όπως τα περισσότερα αντίστοιχα δικαστήρια, όπου η επιλογή μπορεί να λάβει υπόψη και το φόρο του εργασίας και τη διαθεσιμότητα των δικαστών. Πρόκειται για μια ριζική καινοτομία σε σχέση με ένα σύστημα όπου τα μέλη επιλέγουν τους τρεις ε, διαιτητές. Σε πολλές περιπτώσεις έμεσα επιλέγουν τον τρίτο διότι οι δύο επιλεγέντες συμφωνούν επί του τρίτου. Στο σύστημα αυτό τα μέλη δεν θα έχουν επιρροή για το ποιος θα εξετάσει μια συγκεκριμένη υπόθεση. Το θέμα της ανεξαρτησίας των δικαστών είναι ένα άλλο θέμα που ανακύπτει. Πρώτο βήμα είναι η αλλαγή του συστήματος αμοιβών. Δεν θα πληρώνονται από τα μέρη, τα, τους διαδίκους, αλλά από τα μέλη που μετέχουν στη συμφωνία, δηλαδή Ένωση και ΕΠΑ. Το σύστημα που επιλέξαμε για το δικαστήριο αυτό καθευτό αντλεί από μια σειρά άλλων αντίστοιχων οργάνων όπως το αναθεωρητικό όργανο του ΠΟΕ με μηνιαία αντιμισθία για τους ε, δικαστές που θα ανταποκρίνονται στη δουλειά που θα κάνουν. Όλα ωστόσο αυτά θα καταβάλλονται από τα δημόσια ταμεία των δύο πλευρών. Δεν θα υπάρχει δηλαδή κίνητρο ώστε ένας δικαστής να πολλαπλασιάζει τη διαφορές μεταξύ άλλων διότι κατά τη διάρκεια της ε, τοποθέτησής τους δεν μπορεί να δουλέψουν ως ε, δικηγόροι ή σύμβουλοι σε τέτοιες ε, σε επενδυτικές διαφορές. Τώρα, για τον αθεωρητικό όργανο βλέπουμε έξι μέλη όπως σας είπα, πάλι ο ίδια δύο σύστημα, δύο Ευρωπαίοι, δύο Αμερικανοί, δύο Τρίτοι πάλι τυχαία επιλογή των τριών μελών του κατέφεση αυτού οργάνου, του δευτεροβάθμιου οργάνου. Το ίδιο σύστημα απολαβών από τον δημόσιο κορβανά. Δεοντολογία. Η αμεροληψία και η ανεξαρτησία των δικαστών. Ήδη είχαμε διαπραγματευτεί στο ΣΑΙΤΑ, στη Συμφωνία της ε, Σιγκαπούρης, ένα κώδικα δεντολογίας ε, που αντλεί πολλά από την Ένωση Διεθνών Πάνελ. Αυτό θα γίνει δεσμευτικό και στα μέλη των δύο, του πρωτοβάθμιου και του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου. Η εφαρμογή του κώδικα δεν θα αναπόκειται μόνο στους δικαστές, αλλά θα εμπλέκει και τον πρόεδρο του κάθε δικαστηρίου, του πρωτοβάθμιου και του δευτεροβάθμιου. Κατά βάση δηλαδή θα επιλέξουμε μια, έναν τρίτο. Μια εναλλακτική λύση θα είναι ο πρόεδρος του μονίμου διατητικού δικαστηρίου, ο γενικός γραμματέας του ΙΞΙΔ, ή κάποιο άλλο διεθνές όργανο με δικαιοδοτική εντολή και ικανότητα να εξασφαλίσει την, την ε, αμεροληψία και την ακαιρεότητα των μετεχόντων. Έχουμε ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση των διαφορών. Ένα ερώτημα που τέθηκε αφορούσε το ότι οι, τρίτες, οι τρίτοι χρηματοδοτούν μια διαφορά σε ανταλλαγή ε, σε αντάλλαγμα, με αντάλλαγμα το να πάρουν κάτι από την αποζημίωση. Αυτό δεν μπορούμε να το εμποδίσουμε, αλλά μπορούμε να το κάνουμε διάφανο το θέμα, να είναι γνωστό και να γνωρίζει και το δικαστήριο ότι υπάρχουν, ότι υπάρχει χρηματοδότηση τρίτων. Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει είναι ότι είναι σύνθετο και δαπανηρό το σύστημα. Η αρχικοί υπολογισμοί μας που εντάξει δεν ξέρω πόσο αξίζουν αλλά με βάση, δεν έχουμε στοιχεία αλλά με την εικόνα που έχουμε από παλιές διαφορές και από εκτιμήσεις που κάναμε για την Ένωση ανέχεται περίπου στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ ποσό που θεωρήθηκε θεωρείται εύλογο αν το συγκρίνουμε με το τι επιτυγχάνουμε σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία διαφορών που μπορεί να έχουν τεράστιο κόστος. Τώρα, ο πολλαπλασιασμός των μηχανισμών αυτών μπορεί να είναι θέμα. Ένα κομμάτι της συζήτησης αφορά την γενικότερη ανησυχία για την επίλυση τέτοιων διαφορών από πολυμερείς οργανισμούς. Κάτι τέτοιο απαιτεί ένας πολυμερής οργανισμός, απαιτεί πολυμερή συνένεση. Αυτό δεν μπορεί να γίνει άπαξ. Πρέπει να ξεκινήσουμε προσεγγίζοντας ε, χώρες ομοειδεάτες για να διαμορφώσουμε αυτό το consensus για την ε, διαμόρφωση αυτής της ε, ιδέας και στην πρόταση υπάρχει μια μεταβατική ρύθμιση που λέει ότι όταν υπάρξει μια τέτοια πολυμερής, ε, ένα τέτοιο πολυμερές πλαίσιο θα περάσουμε αρμοδιότητα από το διμερές στο πολυμερές. Τώρα, τι σημαίνουν όλα αυτά για τον επενδυτή. Πώς τα βλέπει ένας επενδυτής αυτά. Ακούσαμε ανησυχίες γιατί υπάρχει ευξημενό κόστος, είναι σύνθετο, ο μηχανισμός είναι περίπλοκος. Ένα στοιχείο που προσθέτει, αλλά δεν πρέπει να παραμεριστεί με ύπαρξη της προσφυγής. Το επιπλέον κόστος αξίζει γιατί παρέχει στο όλο σύστημα μεγάλη σταθερότητα. Βεβαίως έχουμε βάλει κάποιες ε, δικλίδες, προθεσμίες, πολλές προθεσμίες, υποχρεωτικές. Αν δείτε οι προθεσμίες πώς, ε, τι, τι θα δώσουν ε, σε σχέση με το ISTS, με την υποθέση στο ISTS, ε, θα δείτε ότι δεν είναι πολύ μεγαλύτερες. Και μην ξεχνάτε ότι το κόστος ε, βαρύνει τα μέρη. Δηλαδή κάθε μέρος πληρώνει το δικό του, το δικό του κόστος και αν χάσει πληρώνει και της άλλης πλευράς. Δηλαδή αν χάσεις το χρόνο του άλλου το πληρώνεις. Υπάρχει μια σειρά δηλαδή στοιχείων που προσπαθούν να αντισταθμίσουν οποιαδήποτε αποδιδόμενη ή καζόμενη δυσαρέσκεια του επενδυτή. Μην ξεχνάτε επίσης ότι αυτός είναι ο τρόπος για να επαναφέρουμε την αξιοπιστία σε ένα μηχανισμό επίλυσης επενδυτικών διαφορών όταν με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε ότι δεν θα υπάρχει μικρότερη προστασία των Αμερικανών επενδυτών στι ΗΠΑ από του επενδυτέ ε, τρίτων χωρών που έχουν παραδοσιακή συμφωνία με το ISTS θα συνεχίσουν να εποφελούνται των βασικών εγγυήσεων που είναι παρόμοιε με αυτέ που εμεί δίνουμε στου επενδυτέ στην Ευρώπη βάσει τη εθνική νομοθεσία και του, των ευρωπαϊκών συνθήκων και η ποιότητα της επίλυσης διαφορών θα βελτιωθεί πάρα πολύ σημαντικά και πάρα πολύ γρήγορα. Εν τέλει δηλαδή υπολογίζουμε ότι αυτό είναι ένα καλό μήνυμα για να τραβήξουμε επενδυτές στην Ευρώπη και να δώσουμε στους ε, αλλοδαπούς επενδυτές επιπλέον εγγυήσεις ότι στην Ευρώπη θα, εξασφα... θα προστατεύονται όχι χειρότερα από Ευρωπαίους ε, επενδυτές και ίσως και καλύτερα. Θα σταματήσω εδώ, είμαι έτοιμος να απαντήσω όπως σας είπα. Φαντάζομαι ότι όλοι την έχετε μάθει απ' έξω την πρόταση, αλλά ε, δεν είμαι βέβαιος ότι μπορώ να απαντήσω σε όλο, οπότε ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων. Αν ε, δεν μπορώ να απαντήσω, θα το σκεφτώ και θα σας απαντήσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Μάουρο και θα ήθελα καταρχάς να δώσω το λόγο στους κοιόδες εισηγητές και μετά να ακούσουμε και τα άλλα μέλη της Επιτροπής. κυρία κυρία <coughs> Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Πετριτσιόνη για την παρέμβασή σα, όπω είπατε, εδώ και μήνε ζητούμε να αντικατασταθεί ο μηχανισμό επίλυση διαφορών με ένα σύστημα που εξασφαλίζει, και αυτό είναι σημαντικό, το δικαίωμα των κρατών να ρυθμίζουν νομοθετικά ό,τι θέλουν. Η νέα πρόταση από ό,τι φαίνεται πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, επαγρυπτούμε ούτως ώστε να γίνονται σεβαστές οι προϋποθέσεις καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων συμφωνίας με τις εταίρους χώρες. Το νέο σύστημα πρέπει να λειτουργήσει ως, μια δημόσια, ως ένα δημόσιο δικαστήριο χωρίς καταχρηστικές ε, προσφυγές. Θέλω να θέσω μια σειρά ερωτημάτων και να ζητήσω κάποιες διευκρινήσεις για το νέο σύστημα. Ποιες είναι οι αντιδράσεις των εταίρων χωρών με τις οποίες ε, συζητούμε αυτή τη στιγμή. Είναι έτοιμες να δεχθούν το νέο σύστημα. Έχετε άτυπες συζητήσεις με τη ΣΥΠΑ για το θέμα αυτό. Άλλη διευκρίνηση. Μπορείτε να μας πείτε τι υποστήριξη μπορεί να έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πρόσβαση στο σύστημα. Μια χρηματοδοτική υποστήριξη προβλέπεται. Επίση, η Κομισιόν συχνά λέει ότι το νέο σύστημα θα, θα εμποδίσει τι καταχρηστικέ προσφυγέ Μπορείτε να μα δώσετε περισσότερα στοιχεία. Τι κριτήρια θα ακολουθήσετε για να κρίνετε κάποια προσφυγή καταχρηστική. Τώρα για το διεθνέ Δικαστήριο Επενδύσεων είπε ότι θα δουλέψετε με άλλε χώρε για την δημιουργία ενό τέτοιου δικαστηρίου. Ποιε είναι οι χώρε που, ξέ, που έδειξαν ήδη το ενδιαφέρον του, Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και τώρα έχω εγώ το λόγο ο συζητητής. Μαύρο. Μου προκάλεσε κάπως έκπληξη. Αλλά και χαρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε τόσο στα σοβαρά την ε, τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μάλιστα την εφήρμοσε ε, σε ό,τι αφορά ε, σημαντικές στιγμές στη διαδικασία το θέμα των ανεξάρτητων δικαστών. Να μην ορίζονται από τους διαδίκους δηλαδή πλέον. Να υπάρχει ένα θεωρητικό σώμα και να είναι διαφανής η διαδικασία. Και πολύ πιο σημαντικό, πιστεύω ότι η απέτηση για μια σαφή αρχή του right to regulate εξασφαλίζεται στο σημείο 2, στο τμήμα 2, σημείο 2 από, του, από τα μέρη ως ε, μία αρχή η οποία διατρέχει όλο το άρθρο και κυρίως σε ό,τι αφορά την αλλαγή της νομοθεσίας να αναφέρεται ρητά ως τμήμα του Right to Regulate 2.2 ότι κάθε επενδύτη φυσικά θα πρέπει να υπολογίσει ότι μπορεί να αλλάξει νομοθεσία κατά τη διάρκεια της επένδυσής του. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η αρχή. Και, και έτσι ορίζονται πλέον και με σαφήνεια διάφορες έως τώρα αντιευκρίνηστες δυνατότητες επένδυσης. Στο 2-3 ότι αυτό περιορίζεται σε καταστάσεις ε, όπου υπάρχει διακριτική μεταχείριση και το θέμα της απατρίωσης 1 ε, στο 3 και στο 2. Διευκρινίζεται λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις ε, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται και πλέον και θα εξαιρούνται και κάποιες περιπτώσεις. Δεν θα υπάρχει τέτοια δυνατότητα πλέον και έτσι ουσιαστικά περιθωριοποιούνται. Εδώ λοιπόν θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. και κάποια ζητήματα τα οποία ήταν ε, απαράδεκτα από το θέμα του κόστους ε, της εκδίκασης και αυτά ρυθμίζονται. Τρία πράγματα θα ήθελα να ρωτήσω ως επερώτηση. Καταρχάς, τι γίνεται με την εφαρμοσιμότητα. Πρόκειται για ένα καινούριο σύστημα. και δεν υπάρχει στους ε, βασικούς κανόνες. Θα πρέπει να γίνει νέα διαπραγμάτευση. Το πώς θα αντιμετωπιστεί. Κατά δεύτερον, στο έγγραφο του Μαΐου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την εθνική δικαιοδοσία υπήρχαν δύο λύσεις, no U-turn και το δεύτερο η πρώτη λύση είναι ότι μπορεί κανείς ε, ε, να ακολουθήσει ένα τρόπο, αλλά δεν μπορεί να τον αλλάξει αυτό στην ε, πορεία. Και το δεύτερο είναι ότι επιλέγουμε εξ αρχής ποια οδό θα ακολουθήσουμε. Θα μπορούσατε να μας επαναφέρετε ποια είναι η αιτιολόγηση, το no U-turn, δηλαδή το ότι δεν κάνουμε στροφή 180 μοιρών, γιατί το ρυθμίζουμε έτσι. Και τρίτον, όπως σας είπα, το κείμενο περιλαμβάνει πολλά θετικά στοιχεία, αλλά δεν βλέπω τίποτα για την υποχρέωση των επενδυτών. Καλά και τα δικαιώματα των, των επενδυτών, αλλά η υποχρέωση τήρησης των ε, κατευθυντηρίων γραμμών του ΩΣΑ του 2011 θα έπρεπε και αυτή να διατυπωθεί. Ευχαριστώ πολύ και τώρα το λόγο έχει. Ευχαριστώ και ευχαριστώ που ήρθατε και να μας εξηγήσετε αυτό το νέο σύστημα και πώς θα λειτουργεί σήμερα και στο μέλλον. Και εγώ ε, είχα αναρωτηθεί ότι θα γίνει με τις χώρες με τις οποίες τώρα διαπραγματευόμαστε και με τις οποίες θα διαπραγματευτούμε στο μέλλον, ε, τι γίνεται δηλαδή με αυτό το δικαστικό σύστημα ε, ISTS. Ε, ήθελα να ξέρω πάντως ποια είναι η θέση του μέσα στο ένομο, στην ένομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς ακριβώς θα λειτουργήσει σε σχέση με την κείμενη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς θα λειτουργήσει το σύστημα κυρίως σε σχέση με την επιλογή των δικαστών. Πέντε θα εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα γίνεται η επιλογή τους και πώς θα μεριμνήσουμε ούτω ώστε να έχουν γνώση και τεχνογνωσία όλων των διαφορετικών νομικών συστημάτων στο ιστορικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Ακόμη και ε, στο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανάμεσα στην Αγγλία και τη Σκωτία, έχουμε ε, σοβαρές διαφορές. Δύο χιλιάδες το μήνα, είπατε θα είναι η αμοιβή του. πρέπει να είναι φθηνότεροι δικαστέ ε, στον κόσμο. Πώς ακριβώς θα ε, χαλιναγωγήσουμε το, το κόστος. Μιλήσατε για 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Ε, ε, ε, θα είναι και μια επιτροπή που θα αναλάβει τους δικαστές και θα μπορεί να αποφασίσει και την αύξηση του αριθμού τους. Πώς μπορούμε να ελέγξουμε αυτήν την επιτροπή. Ευχαριστώ, η Μαρίτια. Σας ευχαριστώ που εξηγήσατε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φυσικά το ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χαίρομαι που βλέπω το ανέδειξε και σε προτεραιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι ε, όλο το πολιτικό φάσμα επανειλημμένα εξέφρασε τις ανησυχίες του για το ESTS όπως υπάρχει σε περίπου 3.000 ε, διμερείς ε, συμφωνίες στον κόσμο για την αμεροληψία, την ανεξαρτησία των δικαστών, το πεδίο ερμοδιοτήτων, ε, την έλλειψη δυνατότητα προσφυγής και το καθεξής. Όλα αυτά, όπως σωστά είπατε, τα καλύψατε και είναι ένα βήμα προς ένα πολύπλευρο σύστημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και απηχώντας και άλλους συναδέλφους, θα ήθελα να ρωτήσω κι εγώ πόσες χώρες εξέφρασαν την υποστήριξή τους για τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα κράτη-μέλη από την άλλη έχουν απαντήσει, ε, θα ζητήσουν να γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στο εθνικό του σύστημα. Υπάρχει τέτοια πρόθεση. Επίσης, οι διεφιστάμενες διμερείς συμφωνίες που ενέχουν αυτόν τον ε, απαρχαιωμένο μηχανισμό ESDS, πώς ακριβώς ε, ε, θα ενσωματώσουν τη νέα πρόταση. Ε, υπάρχει μια τέτοια φιλοδοξία, μετατραπούν σε πλευρά συστήματα, σε πολύπλευρες συμφωνίες ε, εν τέλει. Και πώς θα αποφύγουμε το forum shopping, ε, αν δηλαδή έχουμε ένα, με, ένα διάδικο από που λειτουργεί βάσει μιας διμερούς συμφωνίας θα έχει την επιλογή να διαλέξει ή τη διμερή συμφωνία που εφήρμοζε μέχρι στιγμής ή ε, το πολύπλευρο αυτό νέο σύστημα. Πώς ακριβώς ε, πιστεύει η τη διμερη συμφωνια που εφηρμοζε μεχρι στιγμη η το πολυπλευρο Επιτροπή θα, εφαρμοστεί τον, το σχέδιό της. Και επειδή μιλάμε για το πλαίσιο TTIP, οι εκπρόσωποι της Αμερικανικής κυβέρνησης πώς τοποθετούνται σε σχέση με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ε, μια πολύ έντονη συζήτηση εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σίγουρα την παρακολουθούν και στην Αμερική. Θα ήθελα να ξέρω τι πιστεύουν. Ή οι Καναδοί από την άλλη. Έχετε feedback από αυτούς. Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός για το ε, δικαστήριο που, το ad hoc δικαστήριο που ελπίζουμε και να μην χρειαστεί γιατί μπορεί και να μην προκύψει τέτοια ε, διαφορά θα είναι δηλαδή μια εφημερία, α το πούμε έτσι, δικαστών ε, σε περίπτωση που χρειαστούν. Ποιος θα καλύψει τα έξοδα από πλευράς κράτους μέλους κατά τη διαστολή με ένα προβλεπόμενο και προϋπολογιζόμενο κόστος για ένα μόνιμο ε, δικαστήριο και σε σχέση με την TTIP οι λεπτομέρειες για το δικαστικό μηχανισμό θα ενσωματωθούν στη συμφωνία ή υπάρχει κάποιο σχέδιο α ναι και η τοποθεσία έχει προβλεφθεί κάτι ή θα είναι ένα, ένα περιπλανούμενο δικαστήριο Ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Πετριτσιόνα για τις εξηγήσεις αυτές, οι οποίες ε, ασφαλώς ε, και προβλέθηκαν και στην δημοσιότητα. Πρόκειται για μια συζήτηση την οποία την κάνουμε και ε, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την περνάει παρατηρητή ασφαλώς από το δημόσιο, από την κοινή γνώμη των κρατών Αλλά και στη ΣΥΠΑ φαντάζομαι προβάλλεται. Και πιστεύω λοιπόν ότι είναι σημαντικό και σωστό. Σας ευχαριστώ άλλωστε γι' αυτό. Που το σχέδιο αυτό ήδη δημοσιεύθηκε. Ήδη το σχέδιο δημοσιεύθηκε. Γιατί αυτό συνδέεται και με τη μείωση της αντίστασης του ISDS. Αλλά σε ό,τι αφορά τις εξηγήσεις σας, ότι από τις 150.000 που απόψεις που ακούσαμε, μόνο το 5% είναι υπέρ της συνέχισης του SDS. Τα υπόλοιπα, οι υπόλοιποι είναι υπέρ της ε, διακοπής. Με τη δημόσια συζήτηση λοιπόν ε, διαπιστώνουμε μία απογοήτευση και θα πρέπει να συνεχιστεί η δημόσια συζήτηση. Αλλά θα πρέπει να βηματιστεί λοιπόν αυτή η απογοήτευση. Τρία σημεία θα ήθελα να τονίσω. Ξέρετε ποιες είναι τάσει και οι θέσει τη ομάδα μα. Είμαστε πολύ επικριτικοί, θεωρούμε ότι δεν χρειαζόμαστε ουσιαστικά το ISDS. Να το διευκρινίσω με τρει ερωτήσει λοιπόν αυτό. Καταρχά. το σύστημα ε, για, την, ε, επένδυση, για τις επενδύσεις, ε, έτσι ονομάζεται αυτό, αλλά ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια το ISDS. δεν είναι πραγματικοί δικαστές και στους λέμε δικαστές. Είναι πλούσια άτομα τα οποία είναι νομικοί, με υψηλά προσόντα και πολλές ε, ικανότητες στο θέμα των επενδύσεων και προσβασίας των επενδύσεων, άρθρο 4. Επίσης, τι άλλο προτείνεται και πάλι να υπάρχουν τρεις ε, διαιτητές. Εδώ συνεχίζεται η διαλογική βάση του κειμένου της ε, συμφωνίας, της συνθήκης. Λογικό, αν παραμείνουμε στο σύστημα αυτό. Αλλά όχι βάσει των συνταγμάτων και της νομοθετικής μας βάσης, ούτε στις ΗΠΑ, ούτε των 28 κρατών ε, μελών. Σε ό,τι αφορά δηλαδή ε, συγκεκριμένες, ε, συγκεκριμένους όρους πλαίσιο της επενδύσεις. Και τέλος, θα πρέπει να υπάρχει μια επιτροπή παροχής υπηρεσιών, και επενδύσεων σχετικά με το τι είναι δίκαιο, δίκαιο όρη επενδύσεων. Αλλά τι είναι οι επενδύσει στο 3-3, τι είναι οι επενδύσει, ποιο είναι ο ορισμό. Ε, αυτό, γι' αυτό πάμε το κεφάλι μα. Ε, πολλοί το ερμηνεύουν αυτό ότι ε, θα είναι μια εταιρεία η οποία θα φτιάξει ένα εργοστάσιο και θα δημιουργήσει θέσει εργασία. Αλλά αυτό που προτείνεται στον ορισμό περιλαμβάνει πολλά παραπάνω. Οι επενδύσεις στο εξωτερικό θα πρέπει να προστατεύονται και οι μετοχές ε, και οποιοδήποτε άλλο ε, συμφέρον. Σε ό,τι αφορά την προσδοκία του κέρδους, σε ό,τι αφορά τους φυσικούς πόρους και αυτά πρέπει να προστατευτούν και παραθέτει το αντίστοιχο τμήμα ο μιλητής από, την... από το έγγραφο. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να αντισταθεί κανείς σε κάτι τέτοιο σε επίπεδο διατησίας. Το ερώτημα και την πέντλανε. Τι γίνεται με το θέμα των υποχρεώσεων των πεντετών και αυτά θα πρέπει να αναφέρονται και η δημοσιότητα δηλαδή να μπορεί να αντισταθεί και να υποβάλει ένσταση κατά των αποφάσεων μία εταιρεία. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό. Είναι σημαντικό να μπορούν να τίθενται και τα συμφέροντα των Δήμων και των κοινοτήτων. Σεύρων και Εκουαδόρ. Επί 30 χρόνια συνεχίζεται και εκτελήσεται τη διαφωνία. Δεν έχει ακόμα αποφασιστεί. Πώς γίνεται λοιπόν να υπάρξει περιφερειακή, περιφερειακός σχηματισμός σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Και τώρα ολοκληρώνω το θέμα της, ε, του κόστους. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί ένα στοιχείο της συζήτηση το οποίο συνεχίζεται επί 1,5 έτος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν τελικά πρέπει ο καθένας να πληρώνει από μόνος του τις δαπάνες μια μικρομεσαίας επιχειρήσης οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που υποτίθεται ότι χρησιμοποιούν το TTIP ε, θα είναι σε εκτική θέση, γιατί σε καμία περίπτωση δεν θα μπορέσει να αναλάβει τα δικαστικά έξοδα. Αυτό τι σημαίνει, ότι εκ των προτέρων δημιουργούμε άνισους όρους και νομίζω ότι συνολικά θα έπρεπε να ακολουθήσουμε τη λογική ότι δεν χρειάζεται αυτό το σύστημα εφόσον υπάρχουν τα εθνικά συστήματα για την εκτίκαση διαφορών. Ευχαριστώ Γιάννη. Ευχαριστώ Μπέντ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Ε, δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε, εργαστήκατε σκληρά. Και νομίζω ότι επιδείξατε εκπληκτική δημιουργικότητα κυρίως και στο τίτλο του μηχανισμού, στην ονομασία του μηχανισμού, ε, το οποίο συνιστά μια, αναμφισβήτα μια βελτίωση σε σχέση με το ISTS και εκεί ε, ήσασταν ε, πάρα πολύ δημιουργικοί και πονηροί διότι αλλάξατε την καρδιά του μηχανισμού, δηλαδή ε, τη διαφορά ανάμεσα, τη διεμπλή διαφορών ανάμεσα στους επενδυτές ε, και τα κράτη και δεν φαίνεται αυτό καθόλου στο νέο μηχανισμό. Δεν βλέπουμε δηλαδή ποιοι μετέχουν ε, σε αυτό το νέο μηχανισμό πλέον. Περί τίνος πρόκειται δεν φαίνεται από την επωνυμία του μηχανισμού και πραγματικά όταν το βλέπουμε, ε, ε, όντω πρόκειται για βελτιώσει σε σχέση με το ESDS, αλλά επί τη ουσία δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δηλαδή, πρόκειται για ένα σύστημα ESDS το οποίο ε, έχει ως στόχο να επιλύει τι διαφορέ ανάμεσα στου επενδυτέ και τα κράτη. Απήχοντα τώρα και αυτά που είπε ο Χέλμουτ, την κριτική που σα απίφθηνε, αν κατάλαβα καλά, αυτοί οι δικαστέ θα αμείβονται από αυτόν τον νέο μηχανισμό. Όμως, όταν βλέπουμε ε, τι είδους δικαστές ε, χρειάζεται για αυτή την επιδιαιτησία, ε, αναρωτιόμαστε πώς θα το δεχτούν, πώς θα δεχτούν τόσο χαμηλή αμοιβή, μήπως ε, θα καλύψουν το κενό με διαφορετικό τρόπο, μήπως θα προκύψουν συγκρούσεις συμφερόντων ο δικαστής του πάνελ θα αποφασίσει, θα επιλαμβάνεται τέτοιων ε, περιπτώσεων όπου υπάρχει σίγουρο συμφερόντων και δεν υπάρχει λοιπόν καμία εγγύηση. Και αυτό το νέο φοβερό σλόγγαν, ε, το δικαίωμα της ρύθμισης, ε, αυτό το βλέπουμε πλέον παντού, είναι πάρα πολύ της μόδας και ισχυρίζεται ότι λύνει τα προβλήματα. Επίσης, ε, ε, ουσιαστικά ε, οι διατησίες που γίνονται ποιο αποτέλεσμα έχουν. Δηλαδή, δεν λέμε σε κανένα κράτος μέλος ότι πρέπει να αλλάξετε την νομοθεσία σας. Ποια είναι η ουσία. Χωρίς να τεθεί ένα αμφιβόλο αυτό το δικαίωμα νομοθετικής ρύθμισης ε, του κράτους, ε, παρόλα αυτά δεν συνάδει αυτό που κάνατε με τους στόχους της συνθήκης. Τίποτα περισσότερο. Και άρα, διορθώστε με, αν κάνω λάθος, δεν λύνεται το πρόβλημα της εθνικής νομοθεσίας, δυνάμει της οποίας ο επενδυτής μπορεί να αμφισβητήσει τα εθνικά μέτρα στο βαθμό που είναι επιζήμια για την δραστηριότητά του. Λέτε επίσης ότι δεν είναι πλέον ιδιωτικό το σύστημα και είναι δημόσιο. Ποια είναι η επιχειρηματολογία σας. Μας λέτε ότι στο μέτρο που δημόσιοι φορείς προσλαμβάνουν και επιλέγουν τους δικαστές δεν είναι πλέον ε, ένα σύστημα ιδιωτικού δικαίου. Εγώ πιστεύω ότι εφόσον αυτός ο μηχανισμός επιτρέπει παράκαμψη των αποφάσεων των εθνικών φορέων, των εθνικών θεσμών και ο στόχος του είναι να προστατεύσει τα συμφέροντα ιδιωτικών φορέων, είναι ε, ουσιαστικά ένας μηχανισμός ιδιωτικού δικαίου και όχι δημοσίου δικαίου. Λέτε ότι μπορεί να επιλέξει μια επιχείρηση. Καλά, εξυπακούεται ότι δεν μπορεί να επιλέξει και τους δύο δρόμους. Εντάξει, εάν μια ε, εταιρεία επικαλούμενη άλλα επιχειρήματα και δεν μπορεί να αποταθεί ε, για προβάλλοντας ένα επιχείρημα ε, να αποταθεί σε ένα εθνικό δικαστήριο και προτάσσοντας ένα διαφορετικό επιχείρημα να προσφύγει σε ένα τέτοιο μηχανισμό ISDS, δηλαδή ταυτόχρονα να ακολουθήσει και τους δύο δρόμους, δεν προσθέτει τίποτα στη λύση που επιδιώκουμε εμείς. Ε, δηλαδή δεν μπορεί να έχει και την, ε, το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη το, η, επιχείρηση. Επίσης, ε, τίθεται και ζήτημα εμπιστοσύνης, διότι ε, ωραία κατοχυρώνουμε τα συμφέροντα των επιχειρήσεων, αλλά ούτε οι πολίτες, διότι μόνο οι ιδιώτες, οι επενδυτές μπορούν να ε, προσφύγουν σε ένα τέτοιο δικαστικό όργανο. Όχι οι πολίτες. Και μία ερώτηση στην οποία εξακολουθείτε να μην απαντάτε είναι η θετική διακριτική μεταχείριση που επιφυλάσσεται στους αλλοδαπούς επενδυτές σε, σε αντίθεση με τους εγχώριους επενδυτές. Έχω και άλλα πολλά να σας πω, αλλά θα πω μόνο δύο και φαντάζομαι ότι θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση και θα γίνει το λένε και πιο συγκεκριμένη. Η κυρία Μάλστρομ, από ό,τι ξέρω, επέλεξε τελικά να μην κάνει υποβαλή ένα ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και φαντάζομαι ότι αν κάποιος, ε, παρά, παρότι δεν έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία, παρότι ε, δεν έχει προκύψει νομοθετική ρύθμιση, αποφασίσει κάποιος να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το βρίσκω έξυπνο, διότι θα πρέπει να μπορεί κάποιος να ρωτήσει αν είναι συμβατές αυτές οι ρυθμίσεις με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Και κάτι άλλο, επί του εσείς δεν μας λέτε για ποιο λόγο πρέπει να προκρίνουμε ένα τέτοιο μηχανισμό. Το μόνο που μας λέτε είναι ότι πρέπει να δικαιολογήσουμε αυτά που έχουν γίνει στο παρελθόν, διότι σήμερα δεν υπάρχει καμία μελέτη που να δικαιολογεί και να αποδεικνύει ότι αυτό το σύστημα που είναι καινούριο, που θα πρέπει να ε, συζητήσουμε, που, θα που συνεπάγεται ένα συγκεκριμένο κόστος ε, τι κερδίζουμε σε σχέση με, τους, ε, με τα εθνικά ε, δικαστικά όργανα. Ναι, ακολουθείτε την κατεύθυνση του ψηφίσματο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μα δίνετε τι απαντήσει, πολύ ωραία, αλλά το ζήτημα τη ουσία δεν μα το απαντάτε. Γιατί χρειάζεται αυτό ο νέο μηχανισμό ε, ε, σε σχέση με τα δικαστήρια που υπάρχουν ήδη στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Κύριε Πεγίνη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και εγώ τον ε, προσκεκλημένο μα που παρευρέθηκε σήμερα στην Επιτροπή μα. Όπω θα φαντάζεστε δεν έχω μετακινηθεί στην απόψή μου ότι το ISDS δεν χρειάζεται ως τμήμα του TTIP. Με μεγάλο ενδιαφέρον διάβασα την σας πρόταση και άκουσα και τις κουβέντες που μας είπατε και πραγματικά βλέπω κάποια στοιχεία που έχουν βελτιωθεί αλλά πιο πολλά με ανησυχούν ακόμα. Το ISDS δίνει πιο πολλά κίνητρα στους αλλοδαπούς επενδυτές με άλλα δικαιώματα τα οποία δεν έχουν οι χώροι και αυτό δεν έχει αντιμετωπιστεί. Χαίρομαι που οι οι επενδυτέ θα πρέπει να επιλύουν τι διαφορέ είτε στο εθνικό σύστημα είτε στο καινούργιο ISDS. Αλλά δεν αναφέρεται το γεγονός ότι θα πρέπει να έχουν εξαντλήσει τα εθνικά ένδικα μέσα. Μπορούν να πάνε κατευθείαν στο ISDS, ενώ ο εγχώριος επενδυτής δεν μπορεί να το κάνει αυτό Και αν ε, το εγχώριο συνδικάτο αποφανθεί κατά του επενδυτή, μπορεί να ακολουθήσει με το νέα διαδικασία το δικαστήριο ITS. Ε, άρα θα έχουμε πάλι forum shopping. Δεν έχει πληθεί αυτό το ζήτημα. Επιλέγει καθένα οι αλλοδαποί δηλαδή επενδυτέ ό,τι θέλουν, ό,τι προτιμούν. Και θα ήθελα να ακούσω την άποψή σα για το εξή. Αν ο αλλοδαπό ε, επενδυτή ζητήσει δύο αποζημιώσει, δύο διαφορετικών ειδών αποζημιώσει, μπορεί να προαγάγει την ε, αγωγή του να κάνει αγωγή δηλαδή για με ασφαλιστικά μέτρα να ρωτήσει ή να διαλέξει κάτι άλλο. Και θα πρέπει να προσθέσω ότι δεν ε, αναφέρεται τίποτε για διαδικασίες ε, σε χώρες που δεν είναι μέρη του TTIP. Γιατί να μην είναι μια εταιρεία που να χρησιμοποιήσει τη ρήτρα ISDS που να έχει αλλού τις βασικές της επιχειρήσεις και μόνο ένα μικρό, μια μικρή φυγατρική, στις ΕΙΠΑ. Έχετε απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Δεν το βλέπω αυτό. Και επίσης δεν συμφωνώ με την αισιοδοξία του κυρίου Λάγκη, του Πρόεδρου μας. Δεν βλέπω στην πρόταση. Ρητή και σαφή αναφορά του right to regulate, αυτή την ε, δυνατότητα ρύθμιση. Πώ ε, μα εγγυάται ότι αυτό το ε, όργανο δεν θα μπορέσει να αποφανθεί χωρίς να λάβει υπόψη κάποιους αστικούς νόμους. Και ύστερα οι δικαστές ή οι επιλέγονται από ένα πίνακα. Ποιος μπαίνει σε αυτό το πίνακα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι έχει πληθεί το θέμα Τη μεροληψία υπέρ των επενδύσεων. Αλλά οι επενδυτέ είναι αυτοί που μπορούν να κινήσουν τη διαδικασία και μπορεί οι δικαστέ να είναι υπέρ, να κλείνουν μάλλον υπέρ του επενδυτή. Σας ευχαριστώ πολύ ο πρόεδρο. Οκτώ άλλα άτομα ζητούν το λόγο. Οι συνάδελφοι λοιπόν θα πρέπει να είναι και σύντομη και συνεκτική. Προκειμένου να έχει χρόνο και μόνο να απαντήσει. Jude. Thank you uh, very much. Ευχαριστώ. Αναγνωρίζω την πίεση της Κομισιόν για το θέμα του ISS και την δημόσια αμφισβήτηση του τελευταίου από το κοινό. Εμείς θέλουμε να επιφυλαχθούμε μέχρι να έχουμε μια πλήρη ανάλυση του κειμένου. Μπορεί να φαίνονται βελτιώσεις. Είναι όμως. Νομίζω ότι κάποια θέματα καλύπτονται, αλλά στην ουσία μιλάμε για ένα ξεχωριστό, μια ξεχωριστή ένομη τάξη για τους αλλοδαπούς επενδυτές. Θα ήθελα να ακούσω από την Επιτροπή, την Επιτροπή μας, αν αυτή η μελέτη ασυμβατότητας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τρόπου δικαιοδοσίας θα είναι διαθέσιμη σε εμά. Για τις συγκεκριμένες προτάσεις υπόθηκαν πολλά. Ένα τομέα θέλω να σχολιάσω. Το δικαίωμα νομοθετικής ρύθμισης. Πόσο σφεναρές είναι κατά την αποψή σα οι διατάξεις αυτές. για να μπορέσει να πετύχει ο όρος ε, για την επίτευξη εθνικών ε, στόχων. Ας πούμε, σε περίπτωση που μια κυβέρνηση θέλει να προχωρήσει σε πανεθνικοποίηση κάποιου τομέα, μπορεί να το κάνει. Υπάρχει ο όρος των ε, θεμητών προσδοκιών. Πολλοί δικηγόροι εξέφρασαν επιφυλάξεις για το, τη φράση αυτή. Μια μικρή αλλά πολύ μεγάλη ταυτόχρονα ερώτηση. λέει ότι, αφορά, ότι αυτό αφορά μελλοντικέ συμφωνίες. Για το ΣΑΙΤΑ τι επιπτώσεις έχει. Μάλιστα τον λέει ότι δεν θα το ξεκινήσει, δεν θα το ξαναρχίσει. Κύριε Μενέρη, σας ευχαριστώ και κύριε Πέτρα, σας ευχαριστώ και κύριε Πετριτσιώνα. Έχω ε, κάποια βασικά ερωτήματα να κάνω και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μου απαντήσετε ε, ενδελεχώς και εξειδικευμένως. Το νέο σύστημα ESDS εξακολουθεί να παραμένει ένα σύστημα για την ε, διατησία, για τις διαφωνίες μεταξύ κρατών και επενδυτών. Επενδυτές μπορούν να ε, κάνουν αγωγή κατά το κράτον. Αλλά η Ολλανδία αξιωματοχή της κυβέρνησης τον Απρίλιο του φετινού έτους ανέφεραν ότι οι αλλοδαποί επενδυτές δεν θα έχουν, δεν θα τυχάνουν καλύτερη, σημαντική καλύτερη μεταχείριση σε σχέση με τους εγχώριους επενδυτέ. Αυτό πώς το εξηγείτε στους Ευρωπαίους Υπουργούς. Δεύτερη ερώτηση. Τι ένδικα μέσα παρέχεται στους ε, εγχώριους ε, επενδυτές και εργαζόμενους προκειμένου να προσαγάγουν τους αλλοδαπούς επενδυτές. Τρίτη ερώτηση. Η Επιτροπός Μάλλον Στροεπ επανειλημμένα δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τον Καναδά δεν θέλει να ξανανοίξουν και ότι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει σε περίπτωση που δεν μπει η ρήτρα STS στη ΣΕΤΑ. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα από εταιρείε που μέσω μια θεατρική σε μια άλλη χώρα ξεκινούν ε, ε, μια αγωγή κατά άλλων χωρών ή κατά της δικής τους χώρας. Πώς θα γίνει λοιπόν, τι θα κάνετε προκειμένου οι αμερικανικές εταιρείες να μην περάσουν τον Καναδά για να ξανανοίξουν παλιές υποθέσεις ή να ξαναξεκινήσουν ε, αγωγές κατά της ίδιας τους της χώρας. Τι γίνεται και γιατί δεν είναι καλή δηλαδή η, τα εθνικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των ΗΠΑ Αντιστοιχώς έχετε ε, ε, εντοπίσει τα ελαττώματα, έχετε εντοπίσει τις ατέλειες και γιατί δεν δραστηριοποιούμαστε υπέρ της διόρθωσης αυτών. Και τέλος, έχουμε σε πολλές περιπτώσεις το chilling effect σε ό,τι αφορά την, ε, για παράδειγμα το θέμα της ασφαλτούχου άμμου από, για οδηγία για τα καύσιμα και το καθεξής. Αυτές οι περιπτώσεις θα ανατραπούν, θα αντιστραφούν και μας εγγυάστε ότι το νέο σύστημα επιδητησίας θα εξουδετερώσει αυτό το chilling effect. Ευχαριστώ για την παρουσίαση και την ευκαιρία που έχουμε να συζητήσουμε. Μια διαδικαστική ερώτηση θέλω να θέσω. Η συζήτηση πρέπει να εγκριθεί εδώ ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν και διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ. Υπάρχει μια εγγύηση ότι αυτό που το Κοινοβούλιο θα υποστηρίξει θα γίνει δεκτό από τους διαπραγματευτές. Μετά, για άλλες συμφωνίες που συζητώνται αυτή τη στιγμή θα λειτουργήσει ως μοντέλο που θα εγκριθεί λαμβάνοντας το TTIP ως ε, υπόδειγμα. Δηλαδή, εγώ σίγουρα θέλω να δω περισσότερο, έχω περισσότερο χρόνο για να διαβάσω τις λεπτομέρειες και να καταλάβω το περιεχόμενο, αλλά κάτι που με ανησυχεί εξ αρχής, γιατί το θεωρώ ότι είναι αντιφατικό κάπως, έχει να κάνει με το ότι αυτό που θα διέπει την διαδικασία επίλυση των διαφορών θα είναι κάτι δικαστικό ενώπιον δικαστών, γιατί ακόμα εμένα μου φαίνεται ασαφές το τελευταίο αυτό σημείο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είπατε kurz und präzise, αλλά να ευχαριστήσω παρότι θα είμαι σύντομος και επακριβής στον κύριο Πετριτσιόνε που ήρθε. Διότι πραγματικά είπατε είναι πρωτοφανές να, φε, να δημοσιοποιείτε σχέδιο προτάσεων, αλλά νομίζω ότι είναι καλό, διότι έτσι η πρόταση θα βελτιωθεί. Μετά τις συζητήσεις εδώ σήμερα και μετά τις πληροφορίες που θα πάρουμε από τους εμπλεκόμενους φορείς. Εμείς βεβαίως συζητούμε ένα ευρωπαϊκό κείμενο που θα συμπεριληφθεί στο TTIP αλλά και πάλι θα έχει περισσότερες επιπτώσεις διότι εξετάζουμε ένα μοντέλο παγκοσμίου επίπεδου και αυτό νομίζω ότι θα είναι. Μιλήσατε για πολυμερείς ε, δομές επίλυσης διαφορών και για έναν μηχανισμό μεταβατικό. και πότε θα δημιουργηθεί. Στα πλαίσια αυτά νομίζω ότι θα έπρεπε να εξετάσουμε και την Ευρωπαϊκή, τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε αρκετές ε, ενδοευρωπαϊκές ε, συμβάσεις επίλυση διαφορών που περιλαμβάνουν μηχανισμούς επίλυση διαφορών μεταξύ δυτικών και ανατολικών χωρών. Η ερώτησή μου λοιπόν πηγαίνει προς την ίδια κατεύθυνση με τη Μάρικε αλλά εγώ έχουμε από μια ανατολικοευρωπαϊκή χώρα και, και θα είμαι πιο ε, ε, ανοιχτός από αυτήν την συνάδελφο. Εμείς σκεφτόμαστε το ενδεχόμενο μιας ένδο ευρωπαϊκ... ενός ενδοευρωπαϊκού επενδυτικού δικαστηρίου ή σκέφτεστε την σταδιακή εξάλληψη αυτών των δομών επίλυσης διαφορών στις ε, ενδευρωπαϊκές ε, αντίστοιχες δομές. Και θα δούμε πώς θα λειτουργήσει με το σύστημα με επέκταση των ε, υφιστάμενων θεμάτων για την κοινή αγορά. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που ήδη ακούσαμε. Τέλο πάντων, μπορούμε να χαρούμε τουλάχιστον διότι μετά τι διαβουλεύσει που έγιναν για το SDS ε, κινητοποιήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι περισσότεροι που είχαν απαντήσει ήταν κατά του ISDS και εσεί ε, δεν απαντήσατε λέγοντα ότι δεν θα υπάρξει ISDS, αλλά θα ε, προκύψει ένα τροποποιημένο ISDS για να δούμε αν θα είναι καλοπιστικέ οι αλλαγέ ή ουσιαστικέ. Θα ήθελα να πω ότι παραμένω πεπισμένη στο πλαίσιο της ΕΤΑ και του TTIP δεν είναι απαραίτητος αυτός ο μηχανισμός ε, διότι ούτως ή άλλως υπάρχουν σταθεροί δικαιοδοτικοί μηχανισμοί και για τους επενδυτές και για τα κράτη οπότε δεν χρειάζεται να υπάρξει άλλος τρόπος, ε, άλλος δικαιοδοτικός μηχανισμός. Σε σχέση με τις προτάσεις σας θα ήθελα να υποβάλω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτον, για ποιο λόγο δεν προβλέψατε στο μηχανισμό ότι πρώτα θα πρέπει να εξαντλούνται τα εθνικά ένδικα μέσα προτού ε, προσφύγει κάποιο σε ένα τέτοιο μηχανισμό. Τι μα προτείνεται, να εκκινήσουμε μια διαδικασία στα πλαίσια τη δημόσια ένωμη τάξη και κάποια στιγμή να είναι δυνατόν ε, να ζητήσουμε πάυση αυτή τη εθνική διαδικασία και να προσφύγει κάποιο στη συνέχεια ε, σε αυτόν τον ιδιωτικό μηχανισμό. Συμφωνώ με τον κύριο Ζαντό, πρόκειται για ένα ιδιωτικό δικαιοδοτικό όργανο. Ε, τώρα, όταν μιλάμε για την υποχρέωση αποζημίωσης αναιρείται το δικαίωμα ε, της νομοθετικής ρύθμισης. Όταν κάποιος έχει ρυθμίσει με νομοθετικό τρόπο συνέχεια πρέπει να αποζημιώσει, αναιρεί το ένα το άλλο, ε, είναι προβληματικό. Για τους ε, επενδυτές και τις επενδύσεις, μπορείτε να μας πείτε πώς ακριβώς τους ορίζετε για τη διαμεσολάβηση είναι εντελώς διαφανή ο μηχανισμός δεν θα μπορούσαμε να προβλέψουμε ήδη στο στάδιο της διαμεσολάβησης να υπάρξει διαφάνεια ούτως ώστε να γνωρίζουμε ποιες είναι οι περιπτώσεις ε, που ε, θα ρυθμιστούν ε, από αυτό τον μηχανισμό επίλυσης διαφορά και με ποιο τρόπο ρυθμίζονται. Απέσυραν την αγωγή τους, έκαναν πίσω τα κράτη. Πρέπει να ξέρουμε να υπάρχει διαφάνεια για την ανεξαρτησία των δικαστών. Μας λέτε ότι το μέτρο που όταν εκδικάζουν μια υπόθεση δεν έχουν άλλες εκκρεμείς υποθέσεις ε, θεωρούνται ανεξάρτητοι αμερόληπτοι. Υπάρχει και καραντίνα διότι ε, πέρα από την εκδικασία μιας υπόθεσης μπορεί κάποιος να έχει δικηγορικό γραφείο. Ε, δεν θα πρέπει να βλέπουμε και ποιες υποθέσεις τρέχουν εκεί για να εγγυηθούμε την αμεροληψία των δικαστών. Ε, στη συμφωνία TTIP και ΣΥΤΑ, εγώ πιστεύω και αναλαμβάνω δεν χρειαζόμαστε το ISDS. E ε, αν επιμείνετε, τι θα κάνουμε με τη ΣΕΔΑ, γιατί η κυρία Μάλστον μας είπε ότι δεν πρέπει να αναθεωρήσει τη θέση της. Θα παραμείνει ο όσο έχει. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ο έχουμε καλέσει στην ομάδα μας τους ειδικού για τις διαιτητικά ε, δικαστήρια. Του παρουσιάσαμε λοιπόν την πρόταση την οποία μας παρουσιάσε η κυρία Μάλμστρομ και οι εμπειρογνώμονες αποφάνθηκαν ότι τα εθνικά δικαστήρια εργάζονται πολύ πιο γρήγορα και υποβοτικά από ένα τέτοιο ε, οικοδόμημα. Οι επιχειρήσει, οι οποίε έω τώρα ε, επενδύουν και εξαγάγουν δεν έχουμε να πούμε ότι τα, οι διαδικασίε ε, πρέπει να αντικατασταθούν. Άρα φαντάζομαι ότι υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα και κατεύθυνση στην τρέχουσα πρόταση και στην διατύπωση που ε, κάνει η κυρία Μάλμστρομ ε, για τις δημόσιες συμφέροντα και τα δημοκρατικές αρχές. Υποθέτω ότι για όλα αυτά, πίσω από όλα αυτά κρύβεται πολιτική βούληση. Και τίθεται το ερώτημα επίσης του πώς αντιμετωπίζουν τα πράγματα αυτά οι Αμερικανοί. Και κατά πόσον υποστηρίζουν ένα εύρυθμο σύστημα ISDS. Αν ε, ιδρυθεί λοιπόν ένα νέο θεσμικό σύστημα, πώς μπορούμε να προβλέψουμε ε, τις επιπτώσεις αυτού του νέου θεσμικού οργάνου. Και το θέμα είναι λοιπόν είναι θα είναι ένα το όργανο το οποίο θα λαμβάνει αποφάσεις για οποιαδήποτε χώρα, για όλες τις υποθέσεις και μήπως στην περίπτωση αυτή θα είναι υπερβολικός ο πόρτος επί του οργάνου αυτού ή θα δημιουργηθούν διάφορες ε, διάφορα τέτοια όργανα και πώς θα οργανωθεί αυτό από πλευρά χρόνου. Τι δυνατότητε υπάρχουν, γιατί οι επιχειρήσεις ασφαλώς θα εξαρτώνται από την έκδοση γρήγορα να αποφάσουν για να αποφασίσουν κατά πόσο θα επενδύσουν ή όχι. Άρα το θέμα λοιπόν είναι το κατά πόσο μπορεί να ληφθούν αποφάσει. και αν ιδρυθούν διάφορα δικαστήρια, αναρωτιόμαστε, θα είναι όλα σε μία χώρα ή σε διάφορε χώρε, Γιατί ενδεχομένω κάποια θεσμικά όργανα που είναι μακριά από, κάθε, από κάποια χώρα, ενδεχομένω να μην γνωρίζουν επαρκώς τις τοπικές λεπτομέρειες για να μπορούν να αποφαίνονται. Άλλη ερώτηση. Αν θέλουμε να διασφαλίσουμε και να εξασφαλίσουμε την ανεξαρτησία, αλλά οι υποθέσεις οι οποίες εξετάζονται συνεπάγονται πολύ μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Πώς θα διασφαλίσουμε ότι πραγματικά θα υπάρχει ανεξαρτησία ή μήπως θα γίνει απόπειρα να μπουν και κάποιοι κυβερνητικοί παράγοντες στην απόφαση. Άρα, πάρα πολλά ανοιχτά και κρεμή ερωτήματα πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμα στην ιστορία αυτή. Τελευταίο θέμα. Αξίζει τελική ανάλυση να κάνουμε κάτι πολιτικό πώ, το οποίο από οικονομική άποψη δεν έχει επαρκή αιτιολογία ύπαρξη. Ευχαριστώ, Βίκτορ. Ευχαριστώ. Ε, ξεκινώ ευχαριστώντα τον κύριο Πετρουτσιώνα έκανε μια λεπτομεριακή και πλήρη εξήγηση του νέου συστήματος που απαντά σε μόνιμη πίεση που είχε ασκήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό δείχνει και το ρόλο και τις ικανότητες του Κοινοβουλίου στο θέμα αυτό. Μία ερώτηση. Εξετάζει η Κομισιόν το ενδεχόμενο να δημιουργήσει, να συστήσει αντίστοιχες λύσεις όπως αυτές που προανέφερε και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Αυτό δεν είναι τελικό κείμενο. Μία πρόταση διαπραγματευτικού χαρακτήρα είναι. Το έκανε και την προηγούμενη εβδομάδα η κυρία Μάλστομ. Είναι κομμάτι της διαπραγμάτευση. Το τελικό κείμενο θα εγκριθεί και θα γίνει τμήμα διεθνούς δικαίου. Ωστόσο είμαι πεπισμένη ότι η Ευρώπη θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να εξασφαλίσει ότι η πρόταση θα εγκριθεί στο πλαίσιο που αναφέρεται. Διαπραγματεύσεις τώρα με την Κίνα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο στην Κομισιόν να υπάρξει αντίστοιχη λύση στη διμερή συμφωνία μας με την Κίνα, γνωρίζοντας ότι οι δύο πλευρές, η Ευρώπη και η Κίνα, έχουν τελείως, μα τελείως λέω, ε, διαφορετικά ένομα συστήματα που δημιουργούν αβεβαιότητα και αστάθεια για τους επενδυτές. Είτε επενδύουν στην Κίνα είτε στην Ευρώπη. Εξετάσατε ποια είναι η πιθανή στάση της Κίνας στην πρόταση αυτή. Είναι έτοιμη η Κίνα να συμφωνήσει με την Ευρώπη για να συνδιαμορφώσουν το νέο σύστημα. If... Μια τελευταία παρατήρηση. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο λένε. Ελπίζω να μην, ισχύει, να μην είναι κακή για κάποιους η πρόταση αυτή γιατί είναι καλή. Δεν λέω ότι είναι πολύ καλή. Do answer to our uh, concerns and questions. Πάντως νομίζω η πρότασή σας καλύπτει κάποιες ανησυχίες μας. Ευχαριστώ. Κυρία Φρέντσα, πρόεδρε, ευχαριστώ. Η δουλειά μου διευκολύνθηκε από αυτά που είπαν κάποιοι προορίσαντες συνάδελφοι, ο κ. Σόλτς και ο Ζαντονέ. Νομίζω ότι μπροστά μας έχουμε μία συζήτηση που δεν αναιρεί τους βασικούς λόγους για τους οποίους εμείς ως κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και ως επιτροπές τονίσαμε τον επικίνδυνο χαρακτήρα ενός μηχανισμού όπως αυτού του ESDS. Το, σας θυμίζω εγώ μια δήλωση της κυρίας Μάρστον που είπε ότι δεν υπάρχει καμία άμεση σχέση μεταξύ της αύξησης των επενδύσεων και ενό συστήματος επίλυση διαφορών στο πλαίσιο του TTIP. Αν αυτό συμβαίνει, γιατί πιέζουμε τόσο πολύ το ISDS ε, παρότι φωνάζουν οι πολίτες και διαμαρτύρεται το Κοινοβούλιο. Η πρόταση ελπίζω να δείχνει αλλαγή προσανατολισμού για τα κράτη-μέλη Συνοψίζω πάντως. Ένα πλεονέκτημα. Και άλλο πλεονέκτημα των αλλοδαπών περιδών σε σχέση με τους ντόπιου με τις δόσεις επιχειρήσεις. Βάζουμε δικαστές άτομα που έκαναν εμπορικές διαιτησίες μέχρι τώρα και απλά τους δίνουμε το όνομα δικαστές. Πιστεύω ότι για τους βασικούς λόγους ε, που ανέφερα ότι πρόκειται για ένα και καλυμμένο ISDS και γι' αυτό διατηρούμε τις αντιρρήσεις μας και τις ανησυχίες μας. Η κυρία Σκακέλερ. Σας Ευχαριστώ που ήρθατε και μας παρουσιάσατε αυτή την πρόταση. Είπανε ήδη οι συνάδελφοι ότι υπάρχουν κάποια θετικά ζητήματα, αλλά εμείς οι πράσινοι τα είπε και η Γιάννη, θεωρούμε ότι υπάρχει ένα ε, σοβαρό πρόβλημα, διότι υπάρχει ένα παράλληλο σύστημα που είναι εφαρμοστεί μόνο για τους επενδυτές και δεν λαμβάνουμε υπόψη καθόλου τις υποχρεώσεις που έχουν και αυτοί οι επενδυτές. Αυτό είναι ένα γενικό πρόβλημα, αλλά δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Ούτε και θα επαναλάβω όλες τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Φυσικά περιμένουμε με υπομονησία τις απαντήσεις, αλλά κάτι άλλο που νομίζω δεν αναφέρεται, εκτός αν δεν το άκουσα και που το βρίσκω παράξενο, είναι η αμοιβή των δικαστών είναι προκαθορισμένη, αλλά άμα δείτε τις λεπτομέρειες αναφέρεται ότι υπάρχουν και άλλα τέλη και έξοδα που θα αποζημιώνονται στους δικαστές και τελικά τι είναι 3.000 ε, δολάρια την ημέρα. Δεν είναι και τόσο λίγα τελικά. Αυτή είναι η μερίσια αμοιβή. Μάλλον δεν είναι η μερίσια αμοιβή, είναι τα άλλα έξοδα και οι άλλες αποζημιώσεις που θα προσδιοριστούν στη συνέχεια και φτάνουν στα 3.000 ε, ε, δολάρια. Για το εφετείο αυτό, προτείνεται να ακολουθήσουμε αυτά που προβλέπει στο καταστατικό του ΠΟΕ. Μα αυτό δεν είναι ούτε καν χίλια δολάρια, οπότε ανάμεσα ε, στις αμοιβέ του ε, οργάνου σε πρώτο βαθμό δικαιοδοσία ε, και αυτές του οργάνου σε δεύτερο βαθμό δικαιοδοσία υπάρχει μεγάλη διαφορά. Πώς το εξηγείτε. Επίσης, η αλλοδαποί επενδυτέ που δεν έχουν ουσιαστικέ ε, δραστηριότητε ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο μηχανισμό παρότι μα λέτε ότι δεν θα έχουν. Πού ακριβώ ε, το αναφέρετε αυτό Ρίτα, μπορείτε να μα το εξηγήσετε. Πολλέ ερωτήσει περιμένουμε τι απαντήσει. Τρία λεπτά, ελπίζω να μην μου δώσετε τρία λεπτά για να απαντήσω σε όλα αυτά. δεν αμφιβάλλω ότι θα μπορούσατε και να το κάνετε. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας, όσο θέλετε. Λοιπόν, θα προσπαθήσω ε, στο μέτρο του δυνατόν να ομαδοποιήσω ερωτήσει και θα με χωρέσετε εάν ε, παραβλέψω κάτι που είναι σημαντικό, θα μου το θυμίσετε Όμω είμαι σίγουρο αλλιώ ε, να επανέλθω ήδη μερός να σα δώσω οποιαδήποτε λεπτομέρεια τυχόν παραλείψω. Λοιπόν, για να αρχίσω με το θέμα των τρίτων χωρών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι περισσότερε τρίτες χώρε με τι οποίε ε, διαπραγματευόμαστε μας είπαν ότι ενδιαφέρονται για αυτά που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έχουμε κάνει τέτοιες εξαρτήσεις ενημερωτικές, δηλαδή να μην ε, βασιζόμαστε σε δημοσιεύματα του τύπου. Εμείς προσπαθούμε να εξηγήσουμε τι συμβαίνει στο Κοινοβούλιο, τι συμβαίνει στο Συμβούλιο, ε, ποια είναι τα κίνητρα, ποια είναι η ουσία ε, και η ρίζα των ε, ζητημάτων και το, το διάλογο που γίνεται, ούτω ώστε να προετοιμάσουμε, προλιάνουμε το έδαφος όταν τελικά θα έχουμε μια πρόταση να τους κάνουμε. Για την TTIP η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε συγκεκριμένη πρόταση, έχουμε ένα προσχέδιο. Δεν είμαστε λοιπόν σε θέση να μοιραστούμε αυτό το προσχέδιο με άλλους εταίρους. Εγώ πιστεύω ότι όταν έρθει αυτή η ώρα δεν θα ξαφνιαστούν, διότι Παραδείγματο χάρη, ήμουν την περασμένη εβδομάδα στην Ιαπωνία για διαπραγματεύσει ε, και έδωσα στον ομότιμό μου το προσχέδιο που στο μεταξύ είχε δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του εξήγησα γιατί αυτό και όχι κάποιο άλλο. Και το ίδιο θα κάνουμε και με όλους τους εταίρου μας. Οι συνάδελφοι ήταν στην Κίνα την περασμένη εβδομάδα και σίγουρα το ίδιο έκαναν. Δεν μπορούμε να περιμένουμε σοβαρέ αντιδράσει από πλευράς μέχρι να του δείξουμε ένα πιο τελικό σχέδιο ή μια πρόταση. Προ το παρόν είναι πολύ γενικές, ε, καθόλου ειδικέ οι αντιδράσεις που ε, είχαμε από πλευρά του, ε, Δεν μπορούμε να υπολογίζουμε σε αυτό, αλλά πάντως παρεμφερεί ερωτήματα, παρεμφερεί σε σχέση με αυτά που ακούσαμε από την επιχειρηματική κοινότητα και τα κράτη-μέλη, δηλαδή ποιος είναι ο βαθμός περιπλοκότητας, ποιο είναι το κόστος και ποια είναι η διάρκεια της διαδικασίας. Ε, ε, από πλευράς του Βιετναμ, είναι αναπτυσσόμενη χώρα, λοιπόν οι Βιετναμέζοι Κάτι που μας ξαφνιάζει, λαμβάνοντας υπόψη το πολιτικό και το δικαστικό τους ζήτημα, είχαν πολύ πιο θετική προσέγγιση σε σχέση με άλλους ή, λιγότερο επιφυλακτική. Και μας είπαν, εμείς με το επίπεδο ανάπτυξης που έχουμε μπορούμε να διαχειριστούμε ένα σύστημα που έχει αναπτυχθεί για ανεπτυγμένες χώρες, θεμητό το ερώτημα και τους είπαμε, πως ε, προτιθέμεθα να συζητήσουμε τόσο ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Και το ίδιο και με τους Καναδούς. Τους ε, ενημερώνουμε διαρκώς και περιμένουν από πλευράς μας να εξηγήσουμε καλύτερα τι θέλουμε, τι εννοούμε, ποιοι είναι οι στόχοι μας, ε, τι πιστεύουμε ότι μπορούμε να αποκομίσουμε με ένα τέτοιο μηχανισμό. Και ως συνήθως οι Καναδοί αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτά που συμβαίνουν ανάμεσα στις ΗΠΑ και οποιοδήποτε άλλο εταίρο των ΗΠΑ για προφανείς λόγους. Ε, η, σωστά είπατε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καμία πρόθεση να ε, επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις. Ε, μπορούμε να κάνουμε κάποιες προσαρμογές, αυτό δεν αποκλείεται, αλλά προτού γίνει αυτό, προτού ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τους Καναδούς, θα πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε, ποιος είναι ο στόχος μας. Μετά, τι λείπει και τι είναι τώρα δυνατόν. Έχουμε ένα ολόκληρο φάσμα αναθεωρητικών ε, διατάξεων ε, ε, στην ΣΕΤΑ. θα μπορούσαμε δηλαδή ακόμη και μέσω πρόθεσμα να θεωρήσουμε ότι μπορεί να γίνουν προσαρμογές. Όμως ξαναλέω θα πρέπει να τους εξηγήσουμε τι θέλουμε ε, ποια είναι η πρόθεσή μας και να δούμε ποια είναι η αντίδρασή τους και σε αυτό να βασιστούμε. Λοιπόν, κατά την άσκηση της αναθεώρησης ε, προβλέπεται αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά όχι τώρα ε, να επαναλάβουμε τις διαπραγματεύσεις με το κόστος που αυτό συνεπάγεται. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι η Καναδία πριόρι το απορρίπνει γιατί το αυτό τον μηχανισμό ε, του ε, εφετείου, το είχαμε πρωτοσυζητήσει με ε, τους Καναδούς. Τι είδους τώρα τέτοιο δικαιοδοτικό όργανο θέλουμε, θα πρέπει να το συζητήσουμε μαζί τους όταν έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα του στο παρόν. Τους ενημερώνουμε, αλλά δεν κρίνουμε σκόπιμο να συζητήσουμε σε βάθος μαζί τους προτού γνωρίζουμε και ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που έχουμε δεν είναι η θέση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι προσχέδιο. Πρέπει να περάσει από την διαδικασία. Όμως αυτός ε, ο μορφότυπος που ε, προτείνουμε θα είναι και ο μελλοντικό, ακόμη και για την ε, περίπτωση της Κίνας. Με ρωτήσατε αν θα μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε για τι διαπραγματεύσει με όλε τι χώρε. Δεν το ξέρω για να είμαι ειλικρινή μαζί σα. Δεν μπορώ να σα πω ήδη από τώρα ότι θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το μοντέλο σε όλες τις διαπραγματεύσεις. Πάντως δεν θέλουμε να προδώσουμε τις αρχές ε, στις οποίες βασίζεται αυτό το μοντέλο. Ε, τι αυτή περιπτώσει θα πρέπει να αναθεωρήσουμε το σχέδιο, αλλά προς το παρόν βασιζόμαστε σε αυτά που ξέρουμε, σε στις απόψεις των ε, εταίρων μας όπως τις γνωρίζουμε και δεν θεωρούμε ότι υπάρχει κάποιο ανυπέρβλητο πρόβλημα προς το παρόν. Τώρα το τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων έχω σταματήσει να προσπαθώ να προβλέπω τι θα συμβεί στο μέλλον. Ε, για τη ΣΥΠΑ, επειδή ε, πολλοί ρωτήσατε τι θα γίνει με τη ΣΥΠΑ, η αρχική αντίδραση είναι επιφυλακτική, προσεκτική. Θα ανησυχήσουμε για το επιπρόσθετο κόστος για την επιχειρηματική ε, κοινότητα, για το κόστος, για την περιπλοκότητα της διαδικασίας, για ε, τους επενδυτές που θα έχουν μικρότερη προστασία σε σχέση με αυτό που είχαν κατά νου όταν κάνανε τις επενδύσεις. Όμω, ε, ε, κοιτάξτε και οι ΙΠΑ θέλουν να προστατεύσουν αυτό το δικαίωμα για νομοθετική ρύθμιση, για την ε, ε διαφάνεια, για την... Ε, για τη δέουσα επιμέλεια, όπως και εμείς πιστεύω ότι θα ενδιαφέρονταν να το συζητήσουν μαζί μας και μην ξεχνάμε ότι εκείνοι είναι πρωταθλητές στη διαφάνεια. Πάντως έχουμε στη διάθεσή μας τα στοιχεία για να τους πείσουμε ότι και εφικτό είναι και καλή ιδέα αυτό που προτείνουμε. Δικαίωμα ρύθμισης. Right to regulate. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με αυτό το δικαίωμα. Είναι ένα ζήτημα ε, ένας μηχανισμός επίλυση διαφορών που απορρέει από τα δικαιώματα της συγκεκριμένης ε, συνθήκης και όχι από το εθνικό δικαστικό σύστημα. Σε καμία περίπτωση ε, δεν πρόκειται αυτά τα δικαιοδοτικά όργανα να αποφανθούν για τις εγχώριες νομοθετικές ρυθμίσεις. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αναφέρεται ρήτα. Μόνο για τις διατάξεις της συμφωνίας μπορούν να αποφανθούν και αυτή είναι η βάση οποιαδήποτε απάντηση μπορώ να σας δώσω στα ερωτήματα που μου θέσατε. Γιατί χρειαζόμαστε ένα ιδιαίτερο σύστημα, ειδικό σύστημα, διότι είναι διαφορετικοί οι κανόνες που ισχύουν στις διεθνείς συμφωνίες. Το πιο εύλογο ερώτημα είναι γιατί ε, ο επενδυτής, ένας ιδιωτικός φορέας, έχει τέτοια δικονομικά ε, δικαιώματα, ας πούμε έτσι. Το έχουμε συζητήσει στο παρελθόν. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα καινούριο. Θα ήθελα μόνο να σας υπενθυμίσω ότι για τις ε, ε, ιδιωτικές διαφορές είναι τέτοιες που δεν επαρκούν τα εφιστάμενα συστήματα και πέραν αυτού δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε την ε, την εγκυρότητα των νομοθετικών ρυθμίσεων μιας ε, τρίτης χώρας σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε εμείς να το επηρεάσουμε ούτε να, το, ε, να, αποφανθούμε γι' αυτό. Μπορούμε μόνο να επέμβουμε για τις διατάξεις ε, της, ε, της ε, συμφωνίας. Θα ήθελα να αφήσω αυτό το ζήτημα, διότι δεν έχω κάτι καινούριο να προσθέσω, για να ασχοληθώ με τα καινούργια ερωτήματα. Για την ε, δικαστική βοήθεια ε, για τα... Δεν μπορούμε να το ρυθμίσουμε ε, στη συμφωνία. Είναι ανοιχτό το ζήτημα, δεν έχω απάντηση να σας δώσω. Πάντως πρέπει να είναι χώρια η λύση. Αν θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα που θα βοηθάει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας, τότε αυτό είναι ευρωπαϊκό ζήτημα, θα πρέπει να προβλέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν χρειαζόμαστε κανένα σύστημα που να προστατεύει ή να υποχρεώνει σε κάτι τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, ε, τον ΙΠΑ. Υπάρχουν τα υπέρ και τα κατά. Εμείς τι προσπαθούμε να κάνουμε, να πλουστεύσουμε τον μηχανισμό. Το κόστος σίγουρα θα είναι κατώτερο διότι σε κάθε περίπτωση θα πληρώνονται από τον ε, εθνικό προϋπολογισμό οι δικαστές. Τώρα για τους νομικούς συμβούλους, για τους ε, δικηγόρους είναι άλλο το ζήτημα. Ε, όποιος χάσει θα πληρώσει και τα έξοδα του άλλου. Ναι, αν πάει κάποιος στα δικαστήρια και χάσει, ε, έχει σοβαρό πρόβλημα τότε η επιχείρηση. Ε, εάν ταυτόχρονα μία μικροπιστή επιχείρηση θέλει ε, να προσφύγει στο ε, δικαστήριο τον είπα, τότε μπορεί ε, τα δικαστικά έξοδα, να, τα δικά της, να τα καλύψει η Αμερικανική κυβέρνηση. Αλλά πρέπει να αποδείξει ότι έχει μια ε, επιχειρηματολογία που ευσταθεί. Τώρα για τους νομικούς συμβούλους αυτό θα είναι θέμα της επιχείρησης. Για τις καταχρήσεις και τις κυρώσεις κατά αυτών που προσπαθούν να καταχραστούν το σύστημα. Παραδείγματο χάρη, ε, οι εταιρείε ε, γραμματοκιβώτια δεν μπορούν να προσφύγουν σε αυτόν τον ε, μηχανισμό. Έχουμε διατάξεις που ρητά αποκλείουν αυτήν την περίπτωση που ήδη είδαμε ένα υποκατάστημα ή το Διοικητικό Συμβούλιο κάνει μία επένδυση ε, ταυτόχρονα ενώ ήδη γνωρίζουμε ότι εκκρεμεί ε, μία υπόθεση. Είδαμε στον Φίλιπ Μόρι στο Forum Shopping, όλοι θα έχουν αυτή την περίπτωση κατά νου σίγουρα και ε, ο συνδυασμός διαφόρων στοιχείων μέσα στο μηχανισμό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για να μην είναι δυνατές τέτοιες προσφυγές. Τώρα, το ελαφρώς δυσκολότερο ερώτημα είναι τι συμβαίνει εάν υπάρχει ένα πραγματικό υποκατάστημα σε μια τρίτη χώρα μια θηγατρική. Υπήρχε μια περίπτωση, ε, παραδείγματος χάρη μια ευρωπαϊκή επιχείρηση κατά ε, μιας ε, ε, επαρχίας του Καναδά και τελικά έγινε η προσφυγή από την θηγατρική, την Αμερικανική θηγατρική ε, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας γιατί ε, είχαν γίνει επενδύσεις στον Καναδά από εκείνη την, από εκείνη την θηγατρική ε, που λειτουργούσε ως βασική εταιρεία στη ΣΥΠΑ και ε, εκδικάστηκαν 200 εκατομμύρια σε αυτή την υπόθεση. Έχασε τελικά η εταιρεία. Οι επενδύσεις από τρίτες χώρες είναι κάτι που συμβαίνει δεν ε, κάνουμε διακρίσεις κατά εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της υπηκότητας των μετόχων. Όταν λέμε για genuine business, δηλαδή ουσιαστική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι συμβαίνει αυτό, ε, σημαίνει ότι βάσει της νομοθεσίας πρόκειται για ευρωπαϊκή εταιρεία και δεν βλέπουμε γιατί ε, χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο στη συμφωνία και γιατί οι χώρες μας που επενδύουν στις τρίτες χώρες θα πρέπει να έχουν ε, αντίστοιχη προστασία όπως οι αλλοδαπές που δραστηριοποιούνται εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο και μόνο επειδή η έδρα τους είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα της εφαρμοσιμότητας. Να, ένας λόγος για τον οποίο υπάρχει αναφορά ε, σε, στα awards. Είναι μία διεθνής συμφωνία και η εφαρμοσιμότητα του μηχανισμού ε, βασίζεται στο δημόσιο ε, διεθνές δίκαιο. Τι σημαίνει αυτό. Υπάρχουν κάποιες διεθνείς συμφωνίες που επιτρέπουν να ξεφύγει κάποιος από αυτό το σύστημα και να χρησιμοποιήσει το εγχώριο νομικό σύστημα ε, των ε, βάσει της συνθήκης exit. είναι τεχνικά συστήματα των συμβαλωμένων μερών και αυτό προϋποθέτει ότι ε, το δέχονται ε, τα κράτη-μέλη όπου ζητάτε εσείς να εφαρμοστεί αυτή η σύμβαση και σε κάθε περίπτωση πρόκειται για πλευρή. Για πολυμερή σύμβαση. Δεν είναι, ε, υπάρχει ε, βραχυπρόθεσμη λύση. Με ρώτησαν αν τη σύμβαση έξιτε μπορούμε να τη μετατρέψουμε και να την κάνουμε ένα πολυμερές δικαστήριο. Θα έχουμε 160 μέλη, πρέπει να πείσουμε και 160 χώρες να το κάνουν. Πώς φτιάχνει κάποιος ένα, ένα πολυμερές θεσμικό ε, όργανο. Ξεκινάμε από μονοούσες χώρες. Ε, η Ιαπωνία, Καναδάς, ε, είπα οπωσδήποτε θα δούμε πώς θα αντιδράσει ε, η Κίνα γιατί για τις επενδύσεις ε, είναι πιο προοδευτική σε σχέση με τη στάση που τηρεί σε εμπορικά ζητήματα. Ε, Μία καλή πτυχή είναι ότι προκρίνουν πολυμερείς λύσεις σε σχέση με τις διμερείς Θα δούμε λοιπόν ε, αν έχουμε την κρίση μάζα χωρών ε, και στη συνέχεια ε, θα πρέπει να κάνουμε προτάσεις στον... Όμως αυτό είναι απαραίτητο διότι σε άλλες περιπτώσεις αποτύχαμε έχοντας καταθέσει το σχέδιό μας στον ΟΣΑ και στον ΠΟΕ διότι δεν είχαμε κάνει αυτή την προπαρασκευαστική εργασία. τώρα, στο έγγραφο που μας είχατε στείλει υπήρχαν δύο ε, διαφορετικές λύσεις. Ε, η U-turn στροφή 180 μοίρων, εάν θέλετε, σταματάτε κάποια στιγμή την εγχώρια διαδικασία ε, και ακολουθείτε ε, την διεθνή διαδικασία, προκάνετε τη διεθνή προσφυγή ή εξάντε αποφασίζετε να ακολουθήσετε αυτή τη δεύτερη οδό. Αυτές ήταν οι δύο εναλλακτικέ. Ποια είναι όμως ε, η παρενέργεια της δεύτερης λύσης ότι ε, παρακάμπτεται ή παραγωνίζεται την εθνική διαδικασία. Ε, πώς κάνει κάποιος την επιλογή αν δεν ξέρει στο μέλλον θα μπορέσει να εμπιστευτεί ε, να εθνικό δικαιοδοτικό όργανο και μπορεί να σκεφτεί καλύτερα εκ των προτέρων να αποταθώ σε ένα ε, διεθνή, ε, διεθνές δικαιοδοτικό όργανο και γίνεται η πρωταρχική επιλογή του. Δεν γίνεται όμως να τα έχετε όλα δικά σας, ε, πρέπει να επιλέξετε και το θέμα ποιο είναι τα εθνικά ένδικα μέσα, διότι εξορισμού μπορεί να ε, είναι εφαρμοστέα για τα ίδια ε, περιστατικά, αλλά δεν είναι η ίδια περίπτωση. Δηλαδή, ακόμη και αν έχει την ίδια διατύπωση, ένας ε, διεθνής κανόνας ε, δεν, δεν μπορεί να είναι ίδιος με έναν εθνικό κανόνα. Αυτή η επιλογή δεν έχει καμία ε, σχέση με την επιλογή του Διεθνούς ε, Μηχανισμού ε, Διαθέτησης Διαφορών. Ακόμη και στην Ευρώπη υπάρχει μια σειρά προβλημάτων που έχουν να κάνουν με τη διαδικία των διαφορών σε εμπορικά ζητήματα και σε όταν λάβουμε πόσο ότι έχουμε τέτοιε διαφορέ με χώρε που έχουν ευάλωτα δικαστικά συστήματα σε πολλέ περιπτώσει και που υποχρεώνουν ε, τους επενδυτές να προχωρήσουν πρώτα στην εξάντληση του εθνικού ενδικού μέσου πριν προχωρήσουν στη διεθνή διαφορά ε, θα είναι ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Μπορεί η εθνική νομοθεσία να περιλαμβάνει κάποια ε, δυνατότητα λύσης, αλλά στην πράξη αυτό δεν θα γίνει ποτέ είτε διότι δεν έχουν τη δυνατότητα είτε γιατί στερεί πάρα πολύ το θέμα. το θέμα της υποχρέωσης. Στην ερώτησή σας υπάρχουν δύο παράμετροι. Πρώτον, τι είναι υποχρέωση. Η υποχρέωση του επενδυτή περιλαμβάνει ό,τι αναφέρει η νομοθεσία της χώρας. Όταν επενδύει στην Ευρώπη πρέπει να σέβεσαι την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Τελεία. Η υλοποίηση των αποφάσεων είναι στα χέρια των εθνικών δικαστηρίων, όχι των διεθνών δικαστηρίων. Αυτό ισχύει παντού. Έχουμε την ίδια λογική. Οι διεθνοί κανόνε είναι στα χέρια διεθνού δικαιοδοσία, αλλά το ίδιο επιβάρει να εξασφαλίζουμε ότι η εθνική νομοθεσία θα είναι αποκλειστικά στα χέρια ε, των εθνικών δικαστηρίων. Η υποχρέωση λοιπόν των ε, επενδυτών είναι αυτοί που αποφασίζουν, που αποφασίζουμε εμεί γιατί επενδύουν στη χώρα μα. Το ίδιο ισχύει και για τι επενδύσει επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Αυτό που πετύχαμε με τις επενδυτικές αυτές συμφωνίες είναι ότι οι επενδυτές έχουν ουσιαστική προστασία, ένα επίπεδο ουσιαστικής προστασίας για τα δικαιώματα που, που έχουν συγκρίσιμα με αυτά άλλων επενδυτών. Είτε ημεδαπών είτε αλλοδαπών στην Ευρώπη. Ο λόγος για τον οποίο δεν βλέπετε λοιπόν ε, υποχρέωση των επενδυτών είναι γιατί αυτό είναι μια γενική υποχρέωση προς όλους τους οικονομικά συναλλασσόμενους. Η άλλη παράμετρος είναι κάπως διαφορετικότερη, συνδύεται περισσότερο με το θέμα των συμφωνιών και αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη, καθοδηγητικές γραμμές, αλλά αυτό δεν είναι θέμα επενδυτών, είναι ευρύτερο και δεν έχει να κάνει με την ε, συμπεριφορά λοδαπών επενδυτών στην Ευρώπη αλλά και των δικών μας επενδυτών εκτός Ευρώπης. Υπάρχουν στις συμφωνίες μας ε, συνδέσεις προς την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Πόσο προχωράμε όμως σε αυτόν τον τομέα χωρίς να εξέλθουμε του πλαισίου της παρότρινσης, του εθελούσιου χαρακτήρα και της ε, ε, ε, και της εξάρτησής μας από τις διεθνείς καθηγητήριες γραμμές χωρίς να γίνουν υποχρεωτικές αυτές. Δεν θέλετε να πάμε να τους πούμε, θέλετε να συμφωνήσουμε δεσμευτικούς κανόνες ας πούμε για τα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα. Μπορεί να το θέλουμε αυτό. Θέλουμε να το πούμε όμως. Είναι ανοιχτό το θέμα ακόμα. Δεν είναι ολοκληρωμένο. Πάντως δεν βρίσκεται αυτό στο κεφάλαιο των παιδίσεων και γιατί στην πραγματικότητα είναι εκτός επενδύσεων. Είναι πολύ μεγαλύτερο θέμα. Επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο όχι επενδύει αλλά εμπορεύεται ο κόσμος. Αυτή δεσμοί υπάρχουν ε, σε όλη τη συμφωνία, όχι μόνο στο κομμάτι για τις επενδύσεις. Τώρα το ερώτημα είναι να έχουμε προχωρήσει πολύ ή όχι, είναι ένα θέμα ανοιχτό. Και εγώ επαναλαμβάνω πρώτος ότι είναι ένα δύσκολο θέμα. Δεν έχουμε πείσει την πλειοψηφία των εμπορικών μας εταιρεών να προχωρήσουν όσο θα θέλουμε. Αλλά μετά από 20 χρόνια που ασχολούμαστε με το θέμα αυτό Καταλαβαίνω ότι έχουμε προχωρήσει, πάντως αυτό είναι δικό σας. Ε, επιλογή των δικαστών, όλο αυτό το σύστημα. Καταρχάς, ε, θα σας πρότεινα να δώσετε το κείμενο σε ειδικού για τα δικαστικά ζητήματα στη χώρα σας για να μάθετε πώς γίνονται οι επιλογή, πώς γίνεται η επιλογή, η τοποθέτηση, η εκλογή των δικαστών, η αμοιβή τους, ποιες είναι οι διαδικασίες που έχετε στη χώρα σας. Θα δείτε διαφορές, αλλά και πολλές ομοιότητες. Όταν έρθουμε να συναντήσουμε τις διαφορετικές απόψεις μαζί, θα δείτε ότι αυτό που έχω είναι κάτι που δεν είναι μακριά από ένα δικαιοδοτικό σύστημα που έχουμε. Το ασυμβίβαστο πάντως ε, με, την, με τη δικαιοδική δραστηριότητα ισχύει για όλη την θητεία. Το ερώτημα αν τους πληρώνουμε λίγα όσα πρέπει περισσότερα θα δείξει ο χρόνος. Είδαμε συστήματα όπου οι δικαστές επιλέγονται με αντίστοιχα επίπεδα προσόντων και τα δευτεροβάθμια όργανα που είναι αυτά που κοιτάμε κυρίως, αλλά και άλλα. Το Διεθνές Δικαστήριο, το Μόνιμο Δικαστήριο Διεθνικής Δικαιοσύνης, που δεν διαφέρουν πάρα πολύ μαζικά. Το σύστημα είναι μικρή μηνιαία αντιμισθία για την συμμετοχή τους στο σύστημα. Και η μερίσια αποζημίωση, για το, η μερίσια αμοιβή για τον χρόνο που ασχολούνται με μία υπόθεση που είναι το κύριο κομμάτι της αμοιβή και που κάνει ε, ε, ελκυστικό για αυτούς για να ασχοληθούν με το θέμα αυτό. Που τους οδηγεί δηλαδή στο να επιλέξουν αυτή τη δυνατότητα από το να έχουν μια κερδοφόρα δικηγορική δραστηριότητα. Τα προσόντα που επιλέξαμε αφορούν αυτά που αφορούν τις υποχρεώσεις, μάλλον τις, προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος δικαστή στη χώρα του. Είτε σε μια χώρα της Ένωσης, είτε στη ΣΥΠΑ, είτε σε τέτοια χώρα. Δεν είναι μόνο δικηγόροι. Προσπαθήσαμε να εναρμονίσουμε τους όρους, αλλά δεν απέχουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Προσθέσαμε ε, με ένα επίθετο που να λέει εξαιρετικά νομι, εξαιρετικές νομικές ε, γνώσεις. Θέλουμε να φέρουμε καθηγητές νομικής, δικηγόρους, ε, συμβούλους, νομικούς συμβούλους, όχι μόνο όσους έχουν ασχοληθεί με επενδυτικές διαφορές μόνο στην καριέρα τους. Αν αυτό στην πράξη δεν λειτουργήσει θα πρέπει να το προσαρμόσουμε, αλλά στην πράξη δεν βλέπω λόγους να υποψιαζόμαστε ότι αυτό είναι κόστος του συστήματος όπως σας είπα υπολογίστηκε γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ μισό μισό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ευρωπαϊκό κομμάτι θα πληρώνεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Τώρα, αν θα γίνει δεσμευτικό, ναι, αλλά δεν ε, θα πολλαπλασιαστεί το κόστος ε, μακροπρόθεσμα. Σίγουρα όχι γρήγορα, γιατί δεν επικυρώνεται συμφωνίες ε, μια ανοιχτή, το γνωρίζουμε. Πριν λοιπόν αποκτήσει οικονομικά χαρακτηριστικά, θα πάρει χρόνο, θα δούμε που βρισκόμαστε σε μια πολυμερή συμφωνία. Um, the intra-EU issue. Um, well, more generally, the question of old Α, για τις παλιές συμφωνίες τώρα. Τις διμερείς συμφωνίες. Δεν είναι δυνατόν, να, δεν υπάρχει με τη νέα συμφωνία επιλογή forum shopping. Με την μεταβατική ρύθμιση που εγκρίθηκε η Ευρωπαϊκή Συμφωνία υποκαθιστά τις διμερείς συμφωνίες κρατών της Ένωσης με τρίτες χώρες. Όταν παραμείνει ενισχύ μια διμερής ε, επενδυτική συμφωνία, είναι όταν δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Συμφωνία και το αντίστροφο. Άρα δεν μπορεί να υπάρχει διαφορά με, διένεξη μεταξύ Εθνικής και Ευρωπαϊκής Συμφωνίας. Αν νομίζετε ότι το δικό μας κείμενο είναι πολύ αναχρονιστικό, δείτε μερικές διμερείς συμφωνίες. Αλλά πάντα υπάρχει μια προϊστορία. decision in the e how to deal with And that is progressive replacement e Υπάρχει δυνατότητα πάντως της προοδευτικής υποκατάστασης των εθνικών με τη, των δημερών από την Ευρωπαϊκή Συμφωνία. Κομμάτι-κομμάτι. Αυτό δεν είχε συζητηθεί στο Κοινοβούλιο. Βέβαια το πρόβλημα δεν λύθηκε εν μια νυχτή, αλλά η πρόταση αυτή δεν μπορεί να αλλάξει τις γενικές συμφωνίες. Οι συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών της Ένωσης είναι άλλο θέμα. Αυτό στην πραγματικότητα σε έναν ιδεώδη κόσμο δεν υπάρχει, δεν έπρεπε να υπάρχουν διμερεί συμφωνίε με κράτη με, μεταξύ κρατών μελών της Ένωσης. Κοιτάξτε, βέβαια οι συνάδελφοι στην εσωτερική αγορά δεν συμφωνούν απόλυτα, οπότε αυτά που σας λέω, ε, εγώ τα λέω. Αλλά έχω την εντύπωση ότι κάποια στιγμή το ζήτημα θα αντιμετωπιστεί. Κανονικά, δεν χρειαζόμαστε τις συμφωνίες αυτές. Υπάρχει το δικαστήριο της Ένωσης που λύνει οποιαδήποτε τέτοια ενδοευρωπαϊκή διαφορά. I told you there Α, η θέση, κάτι. Είχα ξεχάσει κάτι και τώρα το θυμήθηκα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το βρούμε, γιατί δεν το είχαμε σκεφτεί μέχρι τώρα. να σας το πω πραγματικά ειλικρινά. Βοστόνη σας αρέσει. Στην ουσία στη Βοστόνη γεννήθηκε ε, το αμερικανικό νομικό σύστημα ή να έχουμε κάτι ε, ένα κινούμενο δικαστήριο. Τώρα μεταξύ Βοστόνη Στρασβούργου μπορεί να είναι λίγο πιο μακριά από τη Στρασβούργου Βρυξελών. Κάπου στη μέση ίσως αν θέλετε, στη μέση του Ατλαντικού. Ισλανδία μια χαρά, Γρυλανδία επίσης. Ο ορισμός της έννοιας επένδυσης. Είναι όντως κρίσιμο το θέμα ο κόσμος χρειάζεται προστασία. Η επένδυση σημαίνει ότι εγώ πάω σε μια χώρα να επενδύσω, μεταφέρω, παίρνω τα, τα λεφτά μου, τη, βάζω σε μια τρίτη χώρα για να κερδίσω εγώ και να κερδίσει και η τοπική οικονομία. Αυτό θα πει επένδυση. Αυτό δεν είναι νομικό. Είναι βασική οικονομική έννοια δεν είναι χτίζω μια, ένα εργοστάσιο. Άλλο το να χτίσω εγώ ένα εργοστάσιο σε μια χώρα και άλλο να... Γιατί να υπάρχει διαφορά μεταξύ του να πάω να χτίσω ένα εργοστάσιο και να επενδύσω σε μια οικονομική δραστηριότητα. Τα ίδια, τις ίδιες πάνες βάζω. Η επένδυση ορίστηκε από εμάς ως η χρήση της ιδιοκτησίας για παραγωγικούς σκοπούς. Τώρα, τι είναι απαλωτρίωση. Η στέρηση της περιουσίας είναι. Αυτός είναι ένας κοινός ορισμός άνω των 200 ετών για το τι σημαίνει απαλωτρίωση. Κάποιο που δεν μπορεί να τηρεί αυτόν τον ορισμό δεν θα τη χάνει προστασία από τη συμφωνία. Αυτό μπορεί να γίνεται μόνο αναπερίπτωση. Το είδαμε σε πάμπολε περιπτώσει. Μόνο περίπτωση μπορεί να κρίνουμε αν κάποιο είναι πραγματικό επενδυτή και αξίζει προστασία ή όχι. Οι δικαστέ θα ευθύνονται, θα έχουν ευθύνη να αποφασίσουν αν ένα κράτος θέλει να πει ότι αυτό δεν είναι πραγματική επένδυση, δεν χρειάζεται να απαντήσω εγώ. Θα τεθεί στο δικαστή. Όπως σε κάθε δικαστήριο θα τίθονται, θα τίθονται θέματα αρμοδιότητας, ε, δικαιώματος παρίστασθε, Ένα άλλο ερώτημα. Οι παράλληλες απαιτήσει βάσει κατασφαλιστικών ε, προσφυγών. Η ασφαλι... Σας διευκρινίζω ότι τα ασφαλιστικά μέτρα που περιλαμβάνονται σε, όλα, σε όλες τις ένομες τάξεις δεν λύνουν την απόφαση αλλά εμποδίζουν να γίνει ανεπανόρθωτη μια κατάσταση που θα οδηγήσει στο να είναι μάταιο το τελικό αποτέλεσμα. Η ασφαλιστική, τα ασφαλιστικά μέτρα λοιπόν είναι παντού ανεξάρτητα από αυτόν που κρίνει επί της ουσίας ο δικαστής. Υπάρχει μια διαφορά. Υπάρχει ένας κίνδυνος, συγκεκριμένες δράσεις να καταστρέψουν ή να αλλάξουν ανεπανόρθωτα το αντικείμενο της διαφοράς. Ο δικαστής λέει σταματάμε και προχωρούμε στην επίλυση επί της ουσίας. Δεν είναι ε, και καλυμμένος τρόπος αντιμετώπισης παράλληλων απαιτήσεων. Περιορίζεται σε κοινέ ε, καταστάσεις που βλέπουμε σε όλα τα ένομα συστήματα. Sorry, I'm finding difficult to read some of my own notes. <laughs> Uh, Δεν καταλαβαίνω και μου. Το θέμα για την ε, απόφαση του δικαστηρίου. Για δύο φορές έχουμε, για, δικαστη... για εμπορικά ζητήματα έχουμε πάει δύο φορές στο δικαστήριο, το 1994 και τώρα έχουμε στραφεί προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ξέρω ότι διαφωνούμε για το κατά πόσο είναι κατάλληλη αυτή η νομική διαδικασία, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για μια διαδικασία συμβατή με το κοινωτικό δίκαιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρόκειται να στραφεί προς το δικαστήριο αν δεν έχει αμφιβολίες. Το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει αμφιβολίες δεν σημαίνει φυσικά ότι απαγορεύεται να έχει κανεί αμφιβολίες. Αλλά σημαίνει ότι η κρίση μας σε αυτή τη ε, φάση, η κρίση της νομικής υπηρεσία μας είναι ότι δεν υπάρχει ασυμβατότητα με το σύστημα του κοινωτικού δικαίου, γιατί μιλάμε για κοινωτικό, δεν μιλάμε για κοινωτικό δίκαιο, μιλάμε για διεθνές δίκαιο εδώ, στην προκειμένη περίπτωση. Και επί της ουσίας είμαι πεπισμένο ότι το ουσιαστικό δικαίωμα που δίνουμε στους ε, αλλοδαπούς επενδυτές με τη συμφωνία αυτή δεν είναι διαφορετικά και σε κάποιες περιπτώσεις είναι ε, υποδέστερα των δικαιωμάτων που χορηγούνται από τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Είμαστε λοιπόν αισιόδοξοι με να κοιτάξω τη σημειώσει μου το θέμα του τι συμβαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόεδρε, αυτό θα σας το αφήσω για σας. Δεν ε, πρόκειται καν να το σχολιάσω. Πρόεδρε, όχι, ξέρω ποια είναι η θέση μου. Για μεσολάβηση. να προσέξουμε. Να μην θέτουμε σε ένα δικαιοδοσία για τα πάντα. Να μην βάζουμε, μην δικαστροποιούμε όλα αυτά τα ζητήματα. Η διαμεσολάβηση υποχρεώνει ουσιαστικά το ένα μέλος να εξετάσει την δυνατότητα φιλικής, ε, φιλικού διακανονισμού. Αυτό δεν είναι ενδικό μέσο. Τίποτα δεν υποχρεώνει την κυβέρνηση του κράτους υποδοχής και τις αρχές να αποδεχτεί τη διαμεσολάβηση. Τίποτα στο σύστημα δεν επιβάλλει ποινέ για τη μη αποδοχή διαμεσολάβηση ή για τη μη χρήση της διαμεσολάβηση καν. Το θέμα είναι πολύ απλά. Κατά πόσον θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα όπου όταν υπάρχει διαφωνία αυτόματα στρεφόμαστε σε 11 μέσα. Αυτό το είδαμε και στον ΠΟΕ Δυστυχώ. και αυτό οδήγησε σε απίστευτο πολλαπλασιασμό των ε, δικαστικών αγωγών. Και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, διαπιστώνουμε ότι πρέπει να επανέλθουμε σε ένα σύστημα φιλικού διακανονισμού. Σε όλα τα ένδικα και νομικά συστήματα υπάρχουν τέτοιες προβλέψεις, τέτοιες ρήτρες και ενθαρρύνεται ακόμα και σε εθνικό επίπεδο η εξοδικαστική, ο εξοδικαστικός ε, διακανονισμός. Το θέμα της διαφάνειας. Άλλο θέμα η διαφάνεια και άλλο θέμα, η διαμεσολάβηση. Αν ε, ένα, ένα μέρος της ε, διαμεσολάβησης είναι κρατικός φορέας και ο αντίκτυπος της διαμεσολάβησης έχει συνέπειες στον εθνικό προϋπολογισμό, θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση δημοσιοποίησης του αποτελέσματος. Η διαφάνεια για την ε, διαφωνία, όπως προβλέπετε εδώ, έχει να κάνει με το ότι το να ξέρουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα δεν φτάνει, γιατί σε κάποιε περιπτώσει χρειαζόμαστε να ξέρουμε και τα νομικά επιχειρήματα και ό,τι συνεπάγονται για την πολιτική και για το θέμα της διαφάνειας της αγωγής. Ένα, μια διευκρίνηση για την... Κυρία Φιωρέντσα. Πότε δεν ε, υποστηρίξαμε ότι δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ της προστασίας των επενδυτών και των ξένων άμεσων επενδύσεων. Είπαμε ότι δεν υπάρχει αυτόματη σύνδεση. Δεν υπάρχει αυτόματο μηχανικό τέτοιο σύνδεσμό. Υπάρχουν πάρα πολλέ έρευνε που υποδεικνύουν ότι υπάρχουν αλληλοσυνδέσει. Όταν υπάρχει καλύτερη προστασία των επενδύσεων, υπάρχουν πιο πολλέ επενδύσεις, πιο σταθερέ επενδύσει. Και πώ πετυχαίνουμε αυτή την προστασία, αυτό είναι άλλο θέμα. Οι διεθνεί συνθήκες και συμβάσει αποτελούν μόνο έναν τρόπο προστασίας. Μπορεί να προστατεύσει κανείς το εθνικό, το, στο εθνικό δίκαιο τη επενδύσεις αυτέ. Εμεί το πιστεύουμε αυτό, αλλά δεν συμφωνούν όλοι οι εταίροι μα. Ούτε με τη ΣΥΠΑ απαραίτητα συμφωνούμε για την προστασία, την σωστή προστασία των αλλοδαπών επενδυτών οι Αμερικανοί φυσικά, άμα του ρωτήσει κανείς, θα σου πούν ότι καλή και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα θέλαμε να υπάρχει καλύτερη προστασία των αναταπών επενδύσεων. Εννοείται. Για το θέμα της ε, σύγκρισης με το κατέθεση όργανο. Δεν είμαι 100% σίγουρος, θα το επαληθεύσω και θα σας αποστείλω και γραπτά ένα πίνακα σύγκρισης. Αλλά αυτό που προβλέπετε για τα μέλη του εφετείου είναι παρόμοια με αυτά που προβλέπονται για το σχετικό όργανο του ΠΟΕ. Η αντιμετώπιση, τα έξι μέλη μάλλον του εφετείου, είτε το γράψουμε στο κείμενο είτε όχι, κατά πάσα πιθανότητα θα έχουν ε, μεγαλύτερη ποσοστό απασχόληση από ότι οι δικαστέ στο δικαστήριο, γιατί είναι μόνο έξι στον αριθμό. Είδαμε τι έχει γίνει και στον ΠΟΕ, αντίστοιχα. Και τα μέλη του εφετείου δεν είναι σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, αλλά αφιερώνουν πολύ σημαντικό χρόνο του χρόνου του, πολύ σημαντικό κομμάτι του χρόνου τους ε, στη δουλειά τους για τις αυξήσεις, ε, για τις επιτροπές που υπάρχουν παντού στις διεθνείς ε, συμφωνίες. Αυτά είναι τα μέρη, ξέρετε, δεν είναι ανεξάρτητα σώματα και αποφασίζονται μέσω συνένεσης. Εμείς είμαστε το μισό της Επιτροπής η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε το μισό όλων αυτών των επιτροπών και οι επιτροπές αυτές δεν κάνουν τίποτα αν δεν συμφωνήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο ισχύει και για το αντίστοιχο, το άλλο μέλος, μέρος. Το πώς διαμορφώνεται η στάση μας στην Επιτροπή αυτή, αυτό εξαρτάται από τους δικούς μας νόμους, τη δική μας νομοθεσία σε ό,τι αφορά λοιπόν τις διεθνείς συμβάσεις. Αυτό εξαρτάται από τις ε, συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα ναι, υπάρχει θέμα αν ξεφύγει από τον έλεγχό μας, αλλά δεν θα ξεφύγει αν δεν το ξέρουμε και αν δεν έχουμε εμεί έλεγχο. Η απόφαση αυτή θα ληφθεί λοιπόν. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το τι θα βγει να πει ο εκπρόσωπος της Ένωσης στην Επιτροπή αυτή. Σύμφωνα με την ε, διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία μας. Υπάρχει λοιπόν έλεγχος. Ελπίζω να μην ξέχασα τίποτα. Τίποτα σημαντικό τουλάχιστον. Μα... Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Πρόεδρο. Ήταν πραγματικά εξαιρετική συζήτηση και οι απαντήσει σα ασφαλώ. Φυσικά είμαστε στην αρχή ακόμα σε ό,τι αφορά την εξέταση της πρότασής σα. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να παραμείνουμε σε επαφή. Σας ευχαριστώ. Gut, liebe Kollegen, Kollegen, dann kommen wir zu Punkt 5. Die Monitoring. Στο 5 να περάσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, παρακολούθηση δραστηριοτήτων των ομάδων. Κύριο Εμπορέλη, έχετε να μα πείτε τίποτα για την Ελβετία. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στι 24 Ιουλίου έγινε η πρώτη, η πρώτη ομάδα δραστηριότητα για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και λήφθησε η απόφαση να επικοινωνηθούμε στην ε, Νορβηγία και στην Ελβετία. Για την ε, Ελβετία, καταρχά. Η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου είναι παλιά, παροχημένη από το 1972 την έχουμε. Και μεταξύ άλλων δεν αναφέρει καθόλου το θέμα της ε, επίλυσης των διαφωνιών. Και επιπλέον υπάρχουν και άλλα προβλήματα γιατί έχουμε πάρα πολλέ διμερεί συμφωνίε και άρα είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουμε θέματα εμπορικά ε, κατά τον τρόπο αυτόν. Και αυτό ασφαλώ αποτελεί και πρόβλημα προ τη διαφάνεια. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι οι κοινοί κανόνε για τι δημόσιε συμβάσει και τον τομέα των υπηρεσιών είναι μάλλον αδύναμοι. Και το θέμα και του ε, ισοτιμία, ε, το ελβετικό φράγκο και η έλλειψη συνταγωνιστικότητα για δυτικού μα ε, παραγωγού. Το ίδιο ισχύει και για την Νορβηγία. Δεν υποστηρίζουν τι κυρώσει κατά τη Ρωσία και παρά το γεγονό ότι υπάρχει η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου, οι εξαγωγέ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και το θέμα της εξαγωγή ε, στο ελβετικό φράγκο, ενώ ουσιαστικά για αυτούς ε, υπάρχει duty free. Για την Νορβηγία τα πράγματα είναι διαφορετικά. Για την Νορβηγία υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα μόνο και αυτό είναι το τέλος για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές ε, ε, ανήσιου κρέατος, βόηου κρέατος και έχουν συζητήσει διάφορα λύσεις, αλλά δεν έχει τελικά αποφασιστεί καμία. Υπάρχουν λοιπόν πολλά προβλήματα και στο εγγύς μέλλον αποφασίσαμε να συγκληθεί και πάλι η ομάδα δραστηριότητας, να συμπεριληφθούν εκπρόσωποι και από τις χώρες αυτές, αλλά και κάποιοι εμπλεκόμενοι φορείς, προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε σε βάθος τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η ομάδα για τη ΣΥΠΑ συναντήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου. για το briefing 13-17 Ιουλίου. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι καινούριο. Δεν υπήρχε κάτι καινούριο μάλλον να αναφέρουμε. Δεν συμφωνηθεί κάτι συγκεκριμένο. Όπως είπε και ο Μάουρο, η Επίτροπος είναι στη ΣΥΠΑ αυτή την εβδομάδα για να κάνει μια συνάντηση για την ε, διαπίστωση το πώς της κατάστασης και το πώς μπορούν να επιταχυνθούν οι διαδικασίε δεδομένου ότι οι ΥΠΑ εξακολουθούν να έχουν την προτεραιότητα για την συμφωνία στον ελληνικό. Η Ιαπωνία, 3 Σεπτεμβρίου. Για την Ιαπωνία έλαβε χώρα στις 3 Σεπτεμβρίου η σχετική συνάντηση θα το συζητήσουμε αυτό. Εκουαδόρ. Ο Χέλμουντ Σόλτ έχει το λόγο. Uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάναμε μια ανταλλαγή απόψεων στις 16 Σεπτεμβρίου, πριν από μια εβδομάδα περίπου, με τους δύο υπουργού ε, εμπορίου, δύο από το Εκουαδόρ και με τον Υπουργό Κοινωνικής Ανάπτυξης, την κυρία Σεσίδε Βακανζόντς. Είχαμε λοιπόν αυτή την πολύ καλή ευκαιρία να συζητήσουμε διάφορες λεπτομέρειες για την Κολομβία και το Περού και την πράξη προσχώρησης. Κάναμε έναν απολογισμό πεπραγμένων για αυτά τα εμπορικά ζητήματα και σε σχέση με τις διάφορες πτυχές του ψηφίσματος προσπαθήσαμε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο κεφάλαιο της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα στην εμπορική συμφωνία καθώς και ε, στον πιθανό αντίκτυπο για τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις σε αυτές τις χώρες. Τονίζω επίσης, για να είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο, πως Ε, αν, ε, ποια είναι η θέση των ε, τριών εξαρμοδίων επιτροπών για το Περού και για το Εκουαδόρ. Πώς θα γίνει αυτή η εύρυθμη προσχώρηση του Εκουαδόρ, διότι ένα χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας μόνο. Και το είπαμε όταν διαπραγματευόμασταν και τη συμφωνία στάνστιλ για τα προβλήματα των γενικευμένων προτιμήσεων GSP και την κατάσταση ε, στο Εκουαδόρ, η πραγματικότητα είναι σκληρότερη και περιπλοκότερη από ό,τι περιμένουμε. Ε, η εξελίξεις ε, στο εκατό σχέση κυρίως με την αντιμετώπιση τη στόχης αλλά και γενικότερα των οικονομικο κοινωνικών και περιβαλλοντικών ε, ζητημάτων. Η καταπολέμηση της απερίμωσης ε, στον Αμαζόνιο, ναι μάλλον της αποψήλωσης των δασών, στον αμαζώνει είναι κάτι άλλο που πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη. που γίνω από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Trade μπορεί να μας ε, ε μιλήσει για τις ημερομηνίε για την προσχώρηση. Πέραν από αυτές τις προπαρασκευαστικές εργασίες ελπίζω να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε και την εφαρμογή της Συμφωνίας για την Προσχώρηση. Το θέμα λοιπόν της χρονικών περιορισμών θα πρέπει να λυθεί υπόψη. Τίσα. 17 Σεπτεμβρίου. Η κυρία Ρέντινγκ δεν είναι εδώ να μας πει τι έγινε. Στο δεύτερο γύρο είμαστε. Δεν άκουσα κάτι ιδιαίτερο και θα τα έχουμε και ένα ψήφισμα για την ΤΙΖΑ, οπότε θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε αυτό το θέμα. Βιετνάμ. 22. Καλά η χώρα η σχετική ε, ομάδα. As you know, thank you, Mr. Όπως ξέρετε, Πρόεδρε, λέει ο κύριο Ζαχαντήλ, οι διαπραγματεύσεις ε, επί της αρχής έχουν ολοκληρωθεί στα τη διάρκεια του καλοκαιριού περιμένουμε το τελικό κείμενο και την υπογραφή της συμφωνίας μέχρι το πέρας του τρέχοντος κατά πάσα πιθανότητα αύριο θα έχουμε συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης μετά από τρεις μήνες αν δεν κάνω λάθος και τότε θα μας ενημερώσουν για την ε, τελική φάση των διαπραγματεύσεων τον Ιούλιο δηλαδή και ελπίζουμε σύντομα να πάρουμε και το τελικό κείμενο. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστούμε. Λέει Λάγκε. Ε, θετικές εξελίξεις. Αυτά για την Επιτροπή Παρακολούθηση και περνάμε τώρα στο σημείο 6. Όχι, συγγνώμη. Πρόεδρε, και η Επιτροπή Παρακολούθησης για την Κίνα, την ξεχάσαμε. Σύντομα θα τα πω. Ήταν ε, πριν το καλοκαίρι. Είμαι στη διάθεση των συναδέλφων αν υπάρχουν ερωτήσεις. Ήταν η 17η σύνοδος που έγινε στις 9 Ιουλίου και στις 14 Ιουλίου συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερωθήκαμε για τα ψηφίσματα τη Συνόδου Υψηλού Επιπέδου. Στη συνέχεια μιλήσαμε για την Τράπεζα Επενδύσεων, ε, στοιχεία σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται για τις επενδύσεις. Δεν έχουν σημειωθεί πολλές αλλαγές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελε να συμπεριλάβει το ρυθμιστικό πλαίσιο και την πρόσβαση στην αγορά, να διευρύνει το πεδίο των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή φαίνεται πως ε, η Κίνα προτιμάει κανονική συμφωνία ελευθερού εμπορίου. Δεν θέλει να διευρύνει αυτή τη στιγμή το πεδίο. Επισήμως δε, δεν, ε, το θέμα της, ε, του καθεστώτος ε, της οικονομίας αγοράς δεν εγγράφεται ποτέ επίσημα στην ημερήσια διάταξη, αλλά σε κάθε συνεδρίαση συζητείται. Και στη συνεδρίαση που είχαμε με τον πρέσβη φέτος, το συζητήσαμε επίσης, αυτό επιθυμεί η Κίνα, εν περιπτώσει, να της χορηγηθεί το καθεστώς. Περιμένουμε μια επίσημη πρόταση, Παντώ σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε η Επιτροπή μας να προετοιμαστεί πολύ καλά για να αντιμετωπίσει αυτό το ενδεχόμενο και θα πρέπει να αποτιμήσει όλες τις ε, πτυχές αυτής της πρότασης. Αυτά δεν θα πω άλλα. Αν έχετε ερωτήσεις, εδώ είμαι. Σας ευχαριστούμε. Δεν υπάρχουν ερωτήσεις, αλλά προφανώς το θέμα του καθεστώτου της οικονομίας αγοράς είναι βασικό. Θα μπει στην ημερήσια διάταξη κάποια στιγμή. Λοιπόν, την άλλη φορά. Μάλλον προχωρούμε στο σημείο 6. ΠΟΕ, Υπουργική Σύνοδος. Μια σύντομη εισαγωγή, σύντομη για το 6. Ξέρετε ότι έχουμε τη σύνοδο στο Ναϊρόμπι το Δεκέμβριο. Θα υπάρξει μια αντιπροσωπεία στη διάσκεψη αυτή για να προωθήσει τις θέσεις μας, για να προωθήσουμε τις θέσεις μας, ετοιμάσαμε ένα ψήφισμα. Οι δύο συμπρόεδροι της ε, Steering Conference του ΠΟΕ εδώ και εγώ, μέχρι τώρα δεν υπάρχει συγκεκριμένο αποτέλεσμα για μια αναθεωρημένη ατζέντα της Ντόχα που θα εγκριθεί στο Ναϊρόμπι, αλλά την περασμένη εβδομάδα αναφέρθηκε ότι υπάρχει πιθανότητα κάποιων εξελίξεων στο Ναϊρόμπι με κάποιες παρατηρήσεις για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, ε, τα αναπτυξιακά αποτελέσματα, κάτι για τη γεωργία και τη βελτίωση της διαφάνειας. Ίσως λοιπόν να υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να υπάρξει πρόοδος στην Υπουργική του Ναϊρόμπι του ΠΟΕ. θα ετοιμάσουμε ένα ψήφισμα που θα τονίζει τη σπουδαιότητα αυτών των πολυμερών προσεγγίσεων πέραν όλων των διμερών που συζητούμε εδώ στην Επιτροπή μας. Αυτά. Ξεκινούμε τις συζητήσεις. Ο συνάδελφος έχει το λόγο. Yeah, <clears throat> Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κ. Στακουλά. Να πω δύο λόγια. Οι άλλοι συνολικά είναι ικανοποιημένοι με το ψήφισμα. Ευχαριστή τους συνθηγητές. Ωστόσο, η ομάδα μου έχει να κάνει κάποιες προτάσεις και σκοπεύουμε να καταθέσουμε τροπολογίες, τις οποίες και ελπίζω ότι θα υποστηρίξετε. Να τις συνοψίσω τις πιο σημαντικές εξ αυτών, εν πάση περιπτώσει. Η Επιτροπή μας ε, υποστηρίζει μία νέα παράγραφο για την ε, πολυμερή εμπορία στον ΠΟΕ ότι για να συνεχίσει να αποτελεί τον αγαγόνια λίθος της ευρωπαϊκής πολιτικής και για να συνεχίσει να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμευμένη στο DDA και να προωθήσει τα συμπεράσματα των 10 της Υπουργικής Συνάντησης για την υποστήριξη του πολυμερού συστήματος για τις ε, πολυμερείς συμφωνίες. Τονίζουμε την ανάγκη να υπάρχει συμβατότητα με τον ΠΟΕ και στο μέλλον. Προκειμένου η διαδικασία να μπει στην, ε, στο σύστημα του ΠΟΕ μόλις τυποποιηθεί η σχετική ευρωπαϊκή, το σχετικό ευρωπαϊκό αίτημα. Έχει αλλάξει πάρα πολύ ο κόσμο. ξέρετε. Εκπληκτικά από το 2001. Οι πρόσφατε συζητήσει στην Γενέβη και στι πρωτεύουσε για το πώ θα συνεχιστούν οι συζητήσεις DDA σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή ατζέντα της Ντόχα καταδεικνύουν ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πραγματικότητες και οι συνθήκες του εμπορικού πλαισίου του σημερινού. Ας μην εστιαστούμε υπερβολικά στο τέλειο και χάσουμε και κάτι καλό. Να έχουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση σχετικά με το τι μπορούμε να συμφωνήσουμε. όλο και πιο πολύ απομακρυνόμαστε από τη φιλοδοξία να πετύχουμε κάτι πολύ φιλόδοξο και πολύ αποτελεσματικό στην Αερόβη. Αλλά θα πρέπει συστηματικά να φροντίσουμε ο διαπραγματεύσει του ΠΟΕ να παραμείνουν κεντρικό στοιχείο της περαιτέρω απελευθέρωσης του παγκόσμιου εμπορίου. Στην παράγραφο 2 σε ό,τι αφορά την ειδική και προνομιακή μεταχείριση, όπως το TTIP. Αυτό είναι εγγενέ στοιχείο της οργάνωσης, αλλά πιστεύουμε ότι είναι κάπως ε, υπερβολική η διατύπωση και δεν βοηθάει σε ό,τι αφορά και τις ε, επιθυμίες της Ινδίας, της Κίνας και άλλων αναπτυσσόμενων χωρών που αποφεύγουν την ευθύνη. Θέλουμε κάπως να αποδυναμώσουμε λοιπόν την ε, διατύπωση, μιας και η παράγραφος 10 καλεί τις αναπτυσσόμενες χώρες να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη, το οποίο πρακτικά τι σημαίνει ότι η ειδική και προνομιακή μεταχείριση μπορεί να καταστεί ομοιόμορφη και αυτόματη. Θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη λοιπόν τι ανάγκε των αναπτυσσόμενων χωρών και των υποανάπτυξη χωρών που είναι σε ανάγκη. Αποφεύγουμε, θα θέλαμε να αποφύγουμε τη λέξη διαφοροποίηση στην παράγραφο 10. Αποτελεί κοκκινή σημαία αυτό για τι αναπτυσσόμενες χώρε. Πολύ καλό το μήνυμα της παραγράφου 10, αλλά α το πούμε χωρί να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη αυτή. Διαφοροποίηση, differentiation. Τα πολλά επίπεδα εξελίξεων η ανάγκε μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών. Σε ό,τι αφορά τις προκλησεις το πραγματικό θέμα δεν είναι να αναπτύξει. αλλά το πως αντιμετωπίζουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες, η Ουγγάντα και οι οι αναπτυσσόμενες χώρες και δεν υπάρχει διαφοροποίηση. Παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε πολύ διαφορετική φάση της ανάπτυξής τους. Ας μην πούμε ότι οι διαφορετικές μεταρρυθμίσεις του ΠΟΕ είναι επιτακτικές. Θα θέλαμε, παρόλα αυτά, να συνεχίσει η βελτίωση της λειτουργίας του ΠΟΕ και της αποτελεσματικότητας του ΠΟΕ για τη Συμφωνία Διευκόλυνσης του Εμπορίου, όχι μόνο γρήγορη εφαρμογή, αλλά και επικύρωση από όλα τα μέλη του ΠΟΕ. Αυτό χρειάζεται. Για να μπει σε εγκαίρωσε το MC10. Και τέλος. Να αναφέρω και ένα πρόβλημα που έχουμε στην παράγραφο 16. Δεν είμαστε υπέρ της δημιουργίας μόνιμης αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με ξεχωριστή γραμματεία για τη σχέση με τον ΠΟΕ. Σύμφωνα με τις κανόνες του κανονισμού, η ΙΝΤΑ εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη και αρμόδια για τις σχέσεις με τον ΠΟΕ. Και θα αργολωθεί η διαδικασία όπως έχει σήμερα. Το να υπάρξει μια μόνιμη αντιπροσωπεία με ξεχωριστό γραφείο θεωρώ ότι θα μείωνε τις αρμοδιότητες που είναι πάρα πολύ σημαντικές τη ΣΥΝΤΑ και της γραμματείας. Και θα συμφωνήσετε όλοι, η δουλειά που κάνει η γραμματεία είναι εξαιρετική. Μια ξεχωριστή μόνιμη αντιπροσωπεία θα απέκλειε τη συμμετοχή των μελών σε άλλες αντιπροσωπείες και σε αποστολές. Ενώ κάποια κοινοβουλευτικά λοιπόν ε, σώματα προσπαθούν να μας πάρουν τις ε, αρμοδιότητες, ας μην ε, βάζουμε τα χέρια μας, να βγάλουμε τα μάτια μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Βίνκλερ, εξ ονόματος του κύριου Σάλβα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, μιλώ εξ ονόματος του συναδέλφου με δύο-τρεις παρατηρήσεις. Είναι η φιλοδοξία του Ναϊρόμπι είναι να υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέσματα. Το Κοινοβούλιο πρόσφατα έδωσε το πράσινο φως στην, συμφωνία, στην εμπορική συμφωνία συστήνοντας το Συμβούλιο ε, την πρόθεση της συμφωνίας. Να συγχαρώ εξ ονόματος του Σιόλου Συγητή στη δουλειά των συναδέλφων και να τονίσω ότι αν θέλουμε να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στην πηγή της. Το, η βιώσιμη ανάπτυξη ε, μπορεί να γίνει μόνο μέσω πολυμερών μηχανισμών όπως ε, η συνθήκη, οι εμπορικές συμφωνίες, οι εμπορικές συμφωνίες. Αυτό είναι αντίστοιχο, ιδίω έντονο τώρα. Βλέπουμε την κρίση της μετανάστευσης που αντιμετωπίζει η Ανατολική Ευρώπη. Φαντάζομαι ότι στο Ναϊρόμπι θα υπάρξουν ε, συζητήσεις για μια σειρά θεμάτων, μείωση των επιδοτήσεων και την υποστήριξη στην γεωργική κρίση, κάτι που προφανώ ε, χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα δεν δέχτηκαν. Αυτά ήθελα να πω εξ του συναδέλφου. Έμα. ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και το σχέδιο που προετοιμάσατε για την Υπουργική του Δεκεμβρίου. Ε, πολύ θετικό είναι ο τόνος και αυτό είναι πολύ καλό γιατί όλοι προσβλέπουμε σε μια θετική απόλυξη στο Ναϊρόμπι. Έχω κάποιες επιφυλάξεις ε, για την παράγραφο 10. Αναφέρομαι στην ειδική και διακριτική διαφοροποιημένη μεταχείριση αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα. Όμως ζητείτε την αντιπροσωπή. Αυτό με ανησυχεί πολύ περισσότερο. Μπορείτε να με διαφωτίσετε. Δεν θα υπάρξει επικάλυψη, δεν θα καλύψει, τη, θα κρύψει το ρόλο, ε, τον υποπτικό ρόλο θα έλεγα που έχει η Επιτροπή μας σε αυτό το πλαίσιο. Πώς θα γίνει, ε, ε, υπάρχει ήδη μόνιμη, αυτή η μόνιμη επιτροπή δεν θα αποτελεί επικάλυψη σχέση με το δικό μας έργο. Ευχαριστώ, Χέλμουτ. Να σας ευχαριστήσω για το κείμενο αυτό. Αποτελεί μια καλή βάση, θεωρώ, για μια επιτυχή εργασία και της Επιτροπής Εμπορίου και του Κοινοβουλίου όμως συνολικά. Και στην επόμενη Υπουργική Συμφωνία και στην Steering Committee στο ε. Υποστηρίζω πολλά από τις προστάσεις. Ε, νομίζω ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ιδιαίτερα και τα θέματα τη ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Προκειμένου να μπορέσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει ουσιαστικά στην ε, πρόθεση των ζητημάτων. Στο σημείο 3 και στο σημείο 4, 7 μπορούμε να προτείνουμε να τοποθετηθούμε πιο εκτενώς στο μνημόνιο της Γενέβης, του Πασκαλαμή που ήταν πολύ εντυπωσιακό πώς διευκρινίζει ότι σήμερα η εμπορική πολιτική δεν μπορεί να είναι μόνο εμπορική πολιτική, αλλά θέμα εντατικών σύνδεσης, εντατικής σύνδεσης με το περιβάλλον, τις αλλαγές του κλίματος, της οικονομίας, της ανάπτυξης. Προς την κατεύθυνση αυτή ενδεχομένω να καταθέσουμε και κάποιες σκέψεις για να διευκρινίσουμε πού βρισκόμαστε και αν ο Έλμαρ Μπρόκος, ο πρόεδρος της εξωτερικών υποθέσεων στην πρώτη συνδρία λοιπόν μετά το καλοκαίρι διαπίστωσε ότι τα, προβλάτα, τα προβλήματα των μεταναστών και των προσφύγων θα πρέπει να το αντιληφθούμε επιτέλους. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι στην πολιτική της ανάπτυξης, στην εξωτερική πολιτική θα πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε επί της αρχή τι πρέπει να αλλάξουμε. Τι έχει να κάνει αυτό με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον ΠΟΕ. Και ως εκ τούτου λοιπόν θα Ήθελα να αμφισβητήσω και κάποιες από τις προτάσεις που έκανε ο συνάδελφος Τακούλα. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να καλύψουμε όλους τους πολιτικούς τομείς και να δούμε πού βρίσκεται σε αυτή τη φάση η εμπορική πολιτική. Στο σημείο 8 θα ήθελα να κάνω και μία αφορά να προτείνω να ελέγξουμε γενικά τι γίνεται, τι συμπεριλαμβάνεται στο ψήφισμα της, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, όπου γνωμοδοτήσαμε για το ρόλο του ΟΗΕ και του συστήματος του ΟΗΕ. Εδώ λοιπόν έχουμε το θέμα του ΠΟΕ, να ελέγξουμε και πολιτικά τι γίνεται, να υπάρχει μια συνοχή, να μην υπάρχουν αντιφάσεις να δούμε λοιπόν την βασική, ε, την, βασική έκθεση. Ένα θέμα το οποίο μου λείπει και θέλω να το αναφέρω είναι ότι στο παρελθόν ε, είχαμε συζητήσει για τη σχέση μεταξύ του παγκόσμιου εμπορίου και των ε, προβλημάτων ισοτιμίας ε, και από πλευρά της Βραζιλίας σε μια ομάδα εργασία προτάστηκε να εξετάσουμε αυτόν το σύνδεσμο. Γιατί έτσι μπορούμε να οικοδομήσουμε και μία γέφυρα με την έκθεση που συζητιέται για την ε, απομείωση του χρέους. Και στο 12 ότι είχατε επαφές με το ICA, με την ΤΙΖΑ, με το ICA. Τι κάνουμε με την πολυμερή διάσταση που έχει τεθεί. Και σε ό,τι αφορά την κυρία Ρέντιν και την Τίζα, θα πρέπει να φροντίσουμε να παραμείνει το εμπόριο σε πολυμερή διάσταση και να μην τα κινηθεί προς την διμερή διάσταση. Κατά άλλα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και να πούμε ότι χαιρόμαστε που μας υποστηρίζουν. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παύλο Κρατσότη. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για αυτό το ψήφισμα και σίγουρα ε, μας το σήμερα στη Γενέβη πηγαίνοντας προς το Ναϊρόμπι. Αλλά τη γνώμη μας η καλύτερη λύση για το Ναϊρόμπι ήταν ε, διαφορετική. Χρειαζόμασταν ένα πιο ολοκληρωμένο πακέτο για να γυρίσουμε τις σελίδα σε σχέση με την DTA και να ασχοληθούμε με άλλα ζητήματα και άλλες προκλήσεις, αλλά δεν είναι αυτό δυνατό. Για την ε, χώρια υποστήριξη και την αμερικανική πρόταση, αναφέρθηκατε και εσείς σε αυτή, ε, είναι ένα δύσκολο ζήτημα, αλλά δυστυχώς δεν θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Ένα μικρό πακέτο, όπως το λέω αυτό, που μπορεί να προκύψει από το Ναϊρόμπι, τι σημαίνει. Θα συμφωνήσουμε πρώτα απ' όλα με όλους σας ότι στην πρώτη υπουργική της Κέννη θα ασχοληθούμε κυρίως με τα αναπτυξιακά ζητήματα και στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Κάποιοι θέλουν να μιλήσουν για την ε, περίφημη differentiation, ε, διαφοροποίηση, άλλοι πάλι θέλουν να αποφύγουν αυτή την κακή λέξη. Στη Γενέβη θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε την ίδια μεταχείριση για την Κίνα ή για μια μικρή αφρικανική χώρα. Από πολιτική σκοπιά πρέπει να τονίσουμε αυτό το θέμα. Εάν τελικά επιλέξουμε αυτό το μικρό πακέτο, τι θα κάνουμε με την πρόσβαση στην αγορά, την εγχώρια στήριξη, το Metic Support. Θα τα αφήσουμε για μεταγενέστερες ε, συνόδους. Δύσκολα μπορούμε να βρούμε λύσεις με τις ίδιες συνταγές που έχουμε ακολουθήσει μέχρι στιγμής. Όπως και να έχει, εν ώψη του Ναϊρόμπι πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με τα υπόλοιπα ζητήματα της Ντόχα, ούτως ώστε στον ΠΟΕ να ε, έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις και να μην αφήσουμε όλα τα καινοτόμα στοιχεία ε, για τις περιφερειακές και για τις πολυμερείς συμφωνίες. Στην παράγραφο 7 του ψηφίσματός σας ε, συμφωνούμε με αυτή την προσέγγιση για την επικύρωση επίσης μάλλον δεν χρειαζόμαστε όλα τα μέλη του ΠΟΕ αλλά τουλάχιστον τα δύο τρίτα για το STT και κάποια μη εμπορικά ζητήματα που αναφέρατε κι εσείς. Υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στα δύο. Υπάρχει μια πρόταση παραδείγματο χάρη αυτή τη στιγμή στη Γενέβη, βάσει της οποίας πρέπει να περιμένουν 12 ε, μήνες ε, οι αναπτυγμένες χώρες ε, προτού επιβάλλουν φυτογενομικά μέτρα σε αναπτυσσόμενες χώρες. Υπάρχουν περιορισμοί ως προς την ανάπτυξη και πώς θα χειριστούμε αυτούς τους περιορισμούς σε σχέση και με το εμπορικό όραμα που έχουμε. Ε, εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό θα έχει την καθοριστική σημασία. Είναι απαραίτητες και διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις Πέρα από αυτές τις μεταρρυθμίσεις θα πρέπει από πολιτική σκοπιά ε, να επανασχεδιάσουμε το σύστημα στον ΠΟΕ για να συνειδητοποιήσουμε και ποιος θα είναι ο ρόλος ε, των ε, αναπτυσσόμενων χωρών. Σας ευχαριστώ και επειδή έχει περάσει και η ώρα δεν θα προσθέσω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Λαγία Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Μία γρήγορη παρατήρηση σε ό,τι αφορά την προσωπία. Αυτό είναι μία διατύπωση η οποία συμπεριλαμβανόταν σε διάφορα παλιά ψηφίσματα. Δεν είναι κάτι καινούριο ιδέα. Και βασίστηκε στην εμπειρία που είχαμε κατά το παρελθόν ότι είχαμε πρόβλημα σε κάποιες περιπτώσεις με τις ε, ad hoc ε, αντιπροσωπείες της Επιτροπής μας να συμμετέχουν στις διαδικασίες του Αυτό τώρα εντάξει μπορεί να μην παραμείνει ως έτοιμα. Ας το σκεφτούμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προθεσμία για τροπολογίες 28 Σεπτεμβρίου. Θα ψηφίσουμε στις 15 Οκτωβρίου. Κανονικά. Σας ευχαριστώ. Και τώρα να περάσουμε στην συνεδρίαση των συντονιστών και κλεισμένων των θυρών. Μόνο συντονιστή γραμματεία, νομική υπηρεσία, υπάλληλοι των ομάδων και επιτρέπεται να συμμετέχουν, να παραβρίσκονται στην αίθουσα και οι βοηθοί των συντονιστών. Δύο λεπτά θα περιμένω για να βγείτε από την αίθουσα οι υπόλοιποι.